Καλημέρα σας λέει η Πρόεδρος. Αρχίζουμε τις εργασίες της ακρόασής μας. Ευχαριστώ όλους όσοι είναι παρόντες. Επίσης τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνεργάστηκαν για να οργανώσουμε τη σημερινή εκδήλωση που είναι μια δημοσία ακρόαση η οποία ξεκίνησε ως συνήθως από πρωτοβουλία των Επιτροπών. Αυτό συμβαίνει με την Επιτροπή της οποίας προεδρεύω. Έχουμε αυτές τις 27 αναφορές, οι οποίες η μία μετά την άλλη υπευλήθησαν και κατέληξαν στα γραφεία μας και με αυτές τις αναφορές ανοίγει ένα καινούργιο παράθυρο, ένα καινούργιο κεφάλαιο στην αντιμετώπιση αυτής της χρηματοοικονομικής κρίσης την οποία αντιμετωπίζουμε. Και αυτές οι αναφορές κατέδειξαν πόσο επιφανειακή ήταν η αντιμετώπιση αυτά τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το βασικό πρόβλημα. Τις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η κρίση των χρηματοοικονομικών αγορών, η κατάρρευση των χρηματιστηρίων, που πηγάζει από τις ΗΠΑ και εμόλυνε τις δικές μας αγορές. Είναι κάτι το οποίο οδήγησε τα θεσμικά όργανα και τις κυβερνήσεις να αντιδράσουν με κάποια μέτρα τιμωρητικά ούτω ώστε να περιορίσουν τα τοξικά προϊόντα και τις αθέμητες πρακτικές. Οπότε το πρώτο θέμα ήταν το πώς θα καταφέρουμε μια σταθερότητα στην οικονομία, πώς θα έχουμε ε, ε, εξυγίανση των ε, προϋπολογισμών, των δημοσιονομικών, αντιμετώπιση του χρέους των χωρών μας, το πώς θα συρρυκνωθούν, θα συγκρατηθούν τα σπρέν σε όλη την Ευρώπη και επίσης προηγήθηκαν και κάποιες ενέργειες όσον αφορά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δηλαδή να δώσουμε οξυγόνο σε αυτές, σε αυτές που είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομίας. Και όλα αυτά ανεφίσαν και έχουν να κάνουν με τη καθημερινή των πολιτών, τα δικαιώματά τους και πρέπει λοιπόν να γίνει σχετική αξιολόγηση και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε επομένως τις ε, αιτίες και όχι να συγκρατούμε τα αποτελέσματα εκεί. γι' αυτό σήμερα μελετούμε τα σχετικά με όλες αυτά τα αρνητικά φαινόμενα όσον αφορά τα αρνητικά μέγεθη της οικονομίας μας και όταν έχουμε μία ματιά επομένως στο τι γίνεται όσον αφορά τη σταθερότητα των δημοσιονομικών είπαμε θα πρέπει να κάνουμε τη σημερινή ακρόαση και θα τη χωρίσουμε σε τρεις άξονες, σε τρία μέρη τη σημερινή ημερίδα. Οπότε θα προσπαθήσουμε να έχουμε αυτή την ενιαία αντιμετώπιση και έτσι να έχουμε μια κριτική ανάλυση και μετά σύνθεση. Και γι' αυτό σας είπα ότι αν μάτια τους οι πολίτες σε σχέση με το τι συνέβη και τι συμβαίνει ακόμα τώρα. Κάτι το οποίο θίγει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και πώς ο έρευνα των δημοσιονομικών έχει θίξει τη δημόσια υγεία, το δικαίωμα στην υγεία, στη σύνταξη των πολιτών, ή στη συνταξιοδότηση. Επίσης, Παραπέρα θα συζητήσουμε το τι πρέπει να κάνουμε, ποιες είναι οι εφικτές, οι δυνατές λύσεις. Να εντός προσοχή μας στις λύσεις έχουν ε, ε ανακύψει τις τελευταίες, ε, τα τελευταία χρόνια την εξαπλίδες μέτρων, την διπλή μέτρων, την ε, τραπεζική εποπτεία Να δούμε συγκεκριμένα τι πετύχαμε με αυτά. Αυτά τα οποία επικαλέστηκαν τα ευρωπαϊκά δεσμικά όργανα, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, σαν απάντηση στην κρίση. Και έτσι θα έχουμε μια καινούρια οικονομική, τραπεζική, δημοσιονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη. Τέλος, να δούμε το πώς επί τη βάση αυτών των ε, αναφορών που ήταν η αφορμή για αυτό το σφορό προβληματισμό να δούμε τι έχουν να πούν ε, κάποιοι ομιλητές, κάποιοι συνάδελφοι που θα λάβουν σήμερα και αυτοί προτείνουν με θάρρος να εξετάσουμε εις βάθος το ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιους δημοσιονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη και εκείνοι προσπαθούν να περιγράψουν το πώς με το άρθρο 48 και γενικότερα πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε τις συνθήκες για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτών των τελευταίων ετών και έτσι να επισημανθεί το ποια μπορεί να είναι η λύση στην κρίση. πώς ευθύνονται οι πολίτες, ε, μπορούμε επομένως να δούμε το πώς μπορούμε να τροπίσουμε τις συνθήκες ούτως ώστε αυτό το υπερεθνικό μόρφωμα η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς μπορεί να αλλάξει. Και αυτό θα κάνουμε. Θα έχουμε αυτή την προσέγγιση και εις βάθος θα τα συζητήσουμε. Και τώρα με αυτή τη συντομή σύγκριση θα προχωρήσουμε πιο συγκεκριμένα στο πρώτο τμήμα της συζήτησής μας που ονομάζεται «Γιατί» και επεξηγούμε σαν υπότιτλο ότι πρόκειται για την οικονομική κρίση και την πολιτική λιτότητα που οδήγησαν σε κοινωνική κρίση στην Ευρώπη και πλέον να υπονομεύσουν τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών. Η Ευρώπη υποφίλει να θεωρεί του πολίτε τη ω πρώτη προτεραιότητα και να καταβάλει προσπάθειε για την ευημερία του. Και ήρθε αμέσω τώρα θα δώσω την σκητάλη στην Αντριάννα Τσερετέλη που εργάζεται για την εφημερίδα Σόλε 24 ώρε. Και την ευχαριστώ που ήρθε. Ehm, Καλή σας μέρα. Είμαι δημοσιογράφος. Παρακολουθώ τα ευρωπαϊκά ζητήματα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχω παρακολουθήσει από το Μάστριχτ τα ευρωπαϊκά ζητήματα και έτσι είδα σιγά σιγά πώς εξελίχθηκε η Ευρώπη. Και πρέπει να σας ομολογήσω ότι τον τελευταίο καιρό με έχει απογοητεύσει η εξέλιξη στα ευρωπαϊκά ζητήματα, εξαιτία της κρίσης βέβαια του ευρώ. Και γιατί με έχει απογοητεύσει, γιατί κατά τη γνώμη μου η κρίση του ευρώ κατά κάποιο τρόπο ήταν κάτι μη αναμενόμενο, δεν το περιμέναμε. Δηλαδή η Ευρώπη δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει μια τέτοια κρίση, δεν είχε προετοιμαστεί καθόλου. Οι κύριοι πρωταγωνιστές ήταν τόσο μπερδεμένοι που δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη στρατηγική. Αντίθετα, εν θερμό αντέδρασαν κατά τη διάρκεια των γεγονότων και μάλιστα καθυστέρησαν και πάρα πολύ να αντιδράσουν. Και το αποτέλεσμα ήταν ε, αντιδράσεις εν πλήρη σύγχυση. Η Γερμανία, για παράδειγμα, που ηγείται στην Ευρώπη δίχως άλλο και είναι από τους ιδρυτές της ε, Οικονομικής Ένωσης, έκανε πολύ σοβαρά σφάλματα πολύ σοβαρά λάθη. Και οι Έλληνες επίσης έκαναν πολύ σοβαρά λάθη γιατί μαγείρεψαν τα στατιστικά τους αποτελέσματα και τώρα που έληξε η περίοδος των παχαίων αγελάδων δεν κατάφεραν να βάλουν τα λογιστικά τους σε τάξη διότι ακριβώς βρέθηκαν σε κρίση. Και υπάρχουν και άλλες χώρες, και η Ιταλία αντίστοιχα. Η κρίση λοιπόν αυτή τι μας έδειξε. Μας έδειξε ότι χώρες οι οποίες ήταν, είχαν πολύ καλά αποτελέσματα όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία για παράδειγμα και αυτές βρεθήκαν στο μάτι του κυκλώνα. Έγιναν σφάλματα λοιπόν τα οποία οδήγησαν τις χώρες αυτές στην κρίση πολύ σοβαρά. Η Ιρλανδία βγήκε από την κρίση κάπως, η Ισπανία όμως όχι ακόμα. Έγιναν λοιπόν σοβαρά λάθη οι διάφορες χώρες βρέθηκαν αντιμέτωπες με φούσκες στα ακίνητα. Άλλες χώρες δεν τήρησαν τα κριτήρια του Μάστριχ, της χρηστής διακυβέρνησης και καμία χώρα δεν ήταν προετοιμασμένη για το ξέσπασμα της κρίσης, με τις συνέπειες βέβαια που γνωρίζουμε. Συνεπώς, σήμερα η Ευρωζώνη μέσα σε πέντε χρόνια, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την Ευρώπη οι πολίτες. Και αυτό είναι η πιο δραματική συνέπεια της κρίσης του ευρώ, κατά τη γνώμη μου, και ο τρόπος με τον οποίο διαχειριστήκαμε την κρίση αυτή. Σήμερα λοιπόν η κρίση αυτή γίνεται και κρίση εμπιστοσύνης, διότι είναι πολύ επιφυλακτικός ο Βορράς απέναντι στον Νότο και ο Νότος απέναντι στον Βορρά. Βλέπουμε δηλαδή να δημιουργείται ένα ρήγμα ανάμεσα στο βορρά και το νότο και να ρωτιόμαστε πώς θα βγούμε από την κρίση. Κάθε φορά λοιπόν που μιλάω για αυτό το ρήγμα, ξέρετε, ήδη όταν φτιάχτηκε η Ευρώπη ξέραμε ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο βορρά και το νότο, αλλά τώρα δεν μιλάμε μόνο για οικονομικό ρήγμα, για οικονομικές διαφορές. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλες διαφορές, πολιτιστικές, πολιτικές, που έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις πάνω στο ευρώ και την Ευρώπη. Αυτή η αλλαγή στην οτροπία ανάμεσα στο Βορρά και το Νότο είναι εκείνη η οποία επιδίνωσε ακόμα περισσότερο την κρίση και έκανε τη διαχείρισή της ακόμα πιο δύσκολη. Κρίση η οποία καταρχήν έπληξε τις μεσογειακές χώρες. Η Γερμανία και άλλες βόρειες χώρες αντέδρασαν και πώς αντέδρασαν θέλοντας να επιβάλλουν κυρώσεις, να τιμωρήσουν τους κακούς θεώρησαν τις χώρες αυτές ένοχες και θέλησαν να τις τιμωρήσουν. Πώς κάνοντάς να υποφέρουν. Έτσι σκέφτηκαν. Και εδώ είναι που έρχεται η διαφορά αυτή στην οτροπία ανάμεσα στους καθολικούς και τους προτεστάντες. Μπορεί να μην σας φαίνεται πολύ σοβαρό, αλλά για μένα είναι μια βασική παράμετρος αυτή, η οποία τάραξε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε επίσης το γεγονός ότι οι βόρειες χώρες, οι οποίες ε, κρίνονται αρνητικά από τις χώρες του Νότου, προσπάθησαν να βάλουν στο ειδόλιο τις χώρες του Νότου. Η κρίση δηλαδή τελικά κατάργησε κάθε ιδέα αλληλεγγύης, κάθε ιδέα βοήθειας προς τους δικούς μας και τελικά καταλήξαμε να θεωρούμε τους άλλους εχθρούς μας. Αυτό έπληξε και την σταθερότητα. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν μιλάμε για μια πραγματική κρίση σε ολόκληρη την Ευρώπη πια. Μια ευρωπαϊκή κρίση. Είπαμε ότι μειώθηκε η εμπιστοσύνη του κόσμου στην Ευρώπη και διαπιστώσαμε ότι οι βόρειες χώρες βάσει μιας εσφαλμένης άποψης και βάσει λαϊκισμού τελικά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν θα έπρεπε εκείνοι να χρηματοδοτούν τα σφάλματα των τεμπέλιδων του Νότου. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά και δεν είναι αλήθεια. Γιατί ο Γερμανός φορολογούμενος, σε κάποιο βαθμό, πάντα χρηματοδοτούσε τα σφάλματα των Ελλήνων καταρχήν. Στο μεταξύ δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός αρρωγής. Ο Γερμανός φορολογούμενος λοιπόν πλήρωσε, αλλά από την άλλη μεριά έπαιρνε επιτόκια πιο ψηλά από αυτά που ίσχυαν στην αγορά. Όλα αυτά βέβαια έχουν τις συνέπειές τους και όταν μιλάμε για εγγυήσει. τι σημαίνει αυτό είναι μια εγγύηση η οποία δεν υποχρεώνει μια χώρα να πληρώσει παρά μόνο εάν πτωχεύσει. Κατά την προεκλογική εκστρατεία στη Γερμανία, ακούσαμε ξανά και ξανά την ίδια ιστορία, ότι οι Γερμανοί ε, βοήθησαν να σωθεί η Ευρώπη. Συνέχισαν να ακούνε ότι είναι θύματα οι Γερμανοί της κακή διαχείρισης των χωρών του Νότου. Κάτι που όπω καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ αρνητικό για την συνύπαρξη Βορρά και Νότου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Νότο πάλι νιώθουν επίση θύματα. Είπα, είναι αλήθεια ότι οι βόρειες χώρες είχαν στο μυαλό τους πώς θα τιμωρήσουν τους κακούς του Νότου, αλλά ούτε και οι χώρες του Νότου δείχνουν την καλύτερη δυνατή θέληση για να προχωρήσουν στις μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες. Μέσα στην παγκοσμιοποίηση, με ένα ενίο νόμισμα, είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε μέτρα για την ανταγωνιστικότητα και για να στηρίζουμε όμως και τα κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία σήμερα πλήττονται τόσο πολύ από την κρίση. Διαπιστώνουμε ότι κάποιες χώρες ίσως δεν αναγνώρισαν αρκετά ότι ο κόσμος άλλαξε και ότι οι εγγυήσει που υπήρχαν στη μεταπολεμική περίοδο αποτελούν πλέον μια εξαίρεση. Δεν είναι πια ο κανόνας. Δεν είναι κάτι που θα διατηρηθεί. Δεδομένου και ότι οι οικονομίες μας μάλιστα δεν είναι σε θέση πια να συνεχίσουν την παραγωγή πόρων και ευημερίε που οδήγησαν σε τόσο καλά κοινωνικά συστήματα που είχαμε μέχρι τώρα. Το αποτέλεσμα λοιπόν της αντιπαράθεσης αυτής, της βίαιης μάλιστα θα έλεγα ανάμεσα στο βορρά και τον νότο, ποια είναι. Πρώτον, ότι τίθεται σε αμφισβήτηση πάρα πολλά δικαιώματα, πάρα πολλές κοινωνικές υπηρεσίες, αμφισβητούνται διάφορες εγγυήσει που είχε ο κόσμος μέχρι τώρα. Η αναφορά ψυχάρη, για παράδειγμα, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έρχεται από την Ελλάδα και συνοψίζει σε μία μόνο φράση τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα. Και είναι από τη στιγμή που η Τρόικα έφτασε στις διάφορες χώρες, από τότε ζητήθηκε και η ευρωπαϊκή βοήθεια. Οπότε τήθηκε το θέμα των συλλογικών συμβάσεων, ελάχιστων μισθών, δημόσιες υπηρεσίες, επιδεινώθηκαν υπηρεσίες υγείας. Όλα αυτά αποτελούν την ε, τρομερή συνέπεια που έχει η κρίση στην Ευρώπη. Η Ευρώπη που θέλει βέβαια να παίξει το ρόλο του καλού Σαμαρίτη ολόκληρο τον κόσμο, στηρίζοντας κοινωνικά δικαιώματα, ε, υποστηρίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. κλπ. Τώρα όμως αναγκάζεται να δράσει διαφορετικά. Και αυτή είναι η πιο θλιβερή σελίδα της ιστορίας που ζούμε, που ζήσαμε και που ζούμε ακόμα. Η κρίση δεν έχει τελειώσει δυστυχώς. Σίγουρα ε, υπήρξαν ε, καθεστώτα που οδήγησαν σε λιτότητα, σε υπερβολική λιτότητα, χωρίς όμως να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλαμε. Γιατί η λιτότητα τι στόχο είχε. Είχε την ε, δημοσιονομική εξυγίανση. Το αποτέλεσμα όμως αυτό δεν ήρθε. Οπότε η κρίση, το έλλειμμα, όλα αυτά επιδεινώνονται τώρα. Οικονομικά λοιπόν είδαμε καταστροφή και κοινωνικά, πολιτιστικά. Η κρίση έπληξε την Ευρώπη τρομερά. Όμως από πλευράς δημοκρατίας επίσης υπήρξε κρίση. Και τι εννοώ με αυτό. Η κρίση αυτή, όλοι το γνωρίζουμε, οδήγησε να φτάσει η Τρόικα στις διάφορες χώρες. Την Τρόικα είναι ε, τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εμπειρογνώμονες, ειδικοί, οι οποίοι κάνουν αυτό που οι κυβερνήσεις δεν είναι σε θέση να κάνουν. Μην ξεχνάμε ότι σε τρία χρόνια κρίση στην Ευρώπη, ξέρουμε ότι 19 πρωθυπουργοί έφυγαν από τις θέσεις τους. Περισσότεροι από τα μέλη της Ευρωζώνης. Η Τρόικα λοιπόν είναι εκείνη η οποία πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Αποφάσεις όμως οι οποίες δεν λαμβάνουν μερικές φορές υπόψη τους την πραγματικότητα που επικρατεί στις διάφορες χώρες. Ποια είναι τα εθνικά συστήματα που είναι διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Άρα στα τυφλά λαμβάνονται οι αποφάσεις αυτές. Έτσι τίθεται πάλι σε αμφισβήτηση η Ευρωπαϊκή Συνένεση, η Ευρωπαϊκή Συμφωνία, αλλά και η ίδια η δομή της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε για την νομιμότητα της τάσης αυτής της Τρόικας, η οποία επειδή θέλει βέβαια την σταθερότητα στην Ευρώπη και για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Νόμισμα, τελικά πλήττει την κοινοβουλευτική κυριαρχία. Είναι αυτή μια εξέλιξη ιδιαίτερα σοβαρή, όπως καταλαβαίνετε, και είναι και ένα τραύμα για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και για την Ευρώπη στο σύνολό της. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει πριν από οτιδήποτε άλλο να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Γιατί αναμφίβολα η τεχνοκρατική Ευρώπη είναι μια Ευρώπη που είναι λιγότερο δημοκρατική. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Είναι το ότι η Ευρώπη πλήττεται από τη γερμανική ηγεμονία. Η Γερμανία η οποία είναι ιδρυτικό μέλος και ο ρόλος της φαίνεται να ενισχύεται στο μέλλον. Για να απλοποιήσουμε κάπως τα πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι φταίει για τον ηγεμονικό αυτό ρόλο που παίζει η Γερμανία. Δεν θα έπρεπε να κάνει το αφεντικό στην Ευρώπη. Η πραγματικότητα όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Όταν έχουμε διαζύγιο, όταν έχουμε χωρισμό σε ένα ζευγάρι, ε, τα πράγματα δεν είναι άσπρα ή μαύρα. Οι ευθύνες δηλαδή είναι και από τις δύο πλευρές. Οπότε η γερμανική ηγεμονία σίγουρα συνδέεται και με το γεγονός ότι δεν είχαν πια συνομιλητές. Η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, πού βρίσκονταν, πού βρίσκονταν οι άλλες μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν ξεκίνησε η κρίση, τι έκαναν οι χώρες αυτές για να προσπαθήσουν να αμβλύνουν κάπως αυτήν την τιμωρητική διάθεση των χωρών του Βορρά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία δεν είναι ότι είναι επιθετική. Όχι, είναι η άμυνα η στάση της. Γιατί φοβάται. Φοβάται τους εταίρους της, φοβάται μήπως τελικά την παρασύρουν μέσα σε μια κρίση η οποία θα κρατήσει πολύ και θα καταλήξει στην πτώχευση του ευρώ, κάτι το οποίο θα είναι μεγάλο χτύπημα και για τη Γερμανία, δεδομένων των εγγυήσεων που έδωσε στην αρχή. Καταλήγοντας, θέλω να σας μεταφέρω το εξής μήνυμα. Σήμερα, μετά τις γερμανικές εκλογές, όπου επανεξελέγει η Μέρκελ, στην Ιταλία και σε άλλες χώρες, εννοείται ότι θα δούμε τι συμμαχίες θα φτιάξει τελικά με τους σοσιαλδημοκράτες ε, ή όχι η Μέρκελ, ελπίζουμε, ή τέλος πάντων πολλοί ελπίζουν ότι η κυρία Μέρκελ θα δείξει ένα άλλο πρόσωπο εφ' εξής. Εγώ όμως είμαι πολύ σκεπτική, διότι διαπιστώνουμε ότι η πολιτική λιτότητας φαίνεται να μειώνεται για συγκεκριμένους λόγους, ίσως γιατί η Γερμανία έχει αντιληφθεί ότι η υπερβολή στη λιτότητα οδηγεί στην αποτυχία και ότι η υπερβολική αυτή λιτότητα θα οδηγήσει στα αντίθετα αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη για τη Γερμανία. Οπότε σιγά σιγά μπορεί να αντιλαμβάνεται η Γερμανία ότι είμαστε στο ίδιο καράβι όλοι. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει αυτό. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω όμως ότι θα αλλάξει και θα φτάσει σε την αντιδιαμετρική στάση η Γερμανία. Την ε, Γερμανία του Κόλ δεν θα την ε, ξαναδούμε με το σχέδιο που υπήρχε τότε για τη βοήθεια στις νότιες χώρες και για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Θα έλεγα ότι η Γερμανία ξεκινάει από την αρχή που λέει ο σωσον εαυτό σωθήτο, ότι ο καθένας δηλαδή θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του μόνος του. Είναι μια αντίδραση ουσίας που φάνηκε κατάφορα κατά τη διάρκεια της κρίσης και νομίζω ότι τη στάση αυτή θα συνεχίσει να την έχει η Γερμανία. Θα θέλει δηλαδή ότι ο καθένας θα πρέπει να φροντίσει να βρει την αξιοπιστία του με την ανταγωνιστικότητα και με τη συμμετοχή στις αγορές. Η εξυγένση των δημοσιονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει εφόσον καθίσουμε στο τραπέζι και συζητήσουμε όλοι για αυτή τη διακυβέρνηση για το ευρώ. Αυτό είναι για μένα πολύ βασικό στόχος. Όμω εξακολουθεί να υπάρχει η κρίση εμπιστοσύνη που σας είπα πριν. Το ρήγμα αυτό, οι διαφορέ ανάμεσα στο βορρά και τον νότο που ξέρουμε ότι υπάρχουν και κάτω από αυτές τις συνθήκες θα είναι δύσκολο να ξεκινήσει ένας διάλογος. Οδηγηθήκαμε στο Σύμφωνο Σταθερότητας, έχουμε τη Συμφωνία των Εξοδιών ε, κλπ. κλπ. Η κρίση όντως οδήγησε σε κάποια αποτελέσματα. Υπήρξε μεταφορά κυριαρχίας από κάποιες χώρες. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θέλουμε να πάμε ακόμα πιο μακριά σε αυτό το στάδιο. Συνεπώς, πρέπει να φτάσουμε στη δημοσιονομική εξυγίανση των χώρων του Νότου, πρέπει να φτάσουμε στη σύγκληση Βορρά-Νότου και μετά να προχωρήσουμε σε νέες μεταρρυθμίσεις. Βέβαια, πρέπει να επιστρέψουν και τα κοινωνικά δικαιώματα στην περίπτωση που έχουμε αυτή την οικονομική ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ. Ο σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσερετέλη, για τις παρατηρήσεις σας για την εισήγηση στην οποία έχετε προβεί ως η πρώτη ομιλήτρια όσον αφορά τις αιτίε του φαινομένου. Και τώρα προχωρούμε στον δεύτερο ομιλητή. Πρόκειται για έναν Ισπανό δημοσιογράφο από την πασίγνωστη εφημερίδα ABC. Ονομάζεται Ενρίκε Σερβέτο. Σε ευχαριστούμε που ήρθες Ενρίκε και σου δίνω ευθύ αμέσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μια που τα εξήγησε τόσο ωραία η Αντριάννα, είναι πάρα πολύ εύκολο τώρα εγώ να λάβω το λόγο γιατί δεν μένουν πάρα πολλά να πει Και θα ήθελα τώρα να εξηγήσω σε όσους δεν είναι Ισπανία το γιατί έχουμε τόσους φορείς, τόσες πρωτοβουλίες, τόση συζήτηση για την κατάσταση που επικρατεί στην Ισπανία. Εν μέρη, γιατί έχουμε κάποιους πάρα πολύ δραστήριους βουλευτές. Εν μέρη βέβαια και γιατί είναι πάρα πολύ οργισμένος ο Ισπανικός λαός. Και όσοι περάσαμε τις διακοπές στη χώρα, γνωρίζουμε, καταλάβαμε ότι η κοινωνία είναι οργισμένη με πολλά. Δεν κατάσταση που επικρατεί με το τι έγινε και τι δεν έγινε. Με την ανεργία που είναι ένα από τα στοιχεία που αφορούν, που αφορούν φυσικά το ότι διάθεση και ο κόσμος δεν έχει δουλειά, όταν δεν πάει πληρώσει τους λογαριασμού του. Όταν η κατάσταση αυτή τέλο πάντων έχει να κάνει με την αισιοδοξία, μιλάμε για 5 εκατομμύρια ενέργου. Δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορούν να πληρώσουν τα στεγαστικά τους δάνεια. Έχουν έρθει εδώ πολλοί φορείς σχετικά με αυτό για να σας τα πούν. Και φυσικά είχαμε και πάρα πολλέ περικοπές για τις υπηρεσίες υγείας. Οπότε, πολλές φορές μπορεί να πει κανείς ότι είναι περισσότερο ψυχολογική παρά πραγματική η, ε, η ατμόσφαιρα αυτή της απεσιοδοξίας, αλλά έτσι έγινε. Βέβαια παρά από αυτή την κακή διάθεση, ε, τη δυσαρέσκεια, είναι υγιής η αντίδραση, αλλά τελικά αιτία είναι το ότι δεν μπορεί η κοινωνία να εντοπίσει ή κυρίως να διαπιστώσει τον ένοχο. Οπότε αναζητάτε ο ένοχος. Τι έγινε. Γιατί μου συμβαίνει αυτό. Οπότε και όντως είναι πολύ εκείνοι που μας μίλησαν στην προηγούμενη ας πούμε ε, στην προηγούμενη ακρόαση που έγινε όσον αφορά αυτές τις ε, μετοχές όσον αφορά το μη εξασφαλισμένο χρέος δεν υπάρχει πια στήριξη των ε, τραπεζών που καταβάλει προσπάθεια η χώρα. Ξέρουν τα χρέη και αλλά δεν μπορεί η κοινωνία να διπιστώσει ποιο είναι ο ένοχο, σε ποιον απευθυνθούν για την επίλυση των ε, προβλημάτων. Σε αυτό σα εξηγώ τώρα. Πώ βλέπει τα πράγματα ο κόσμο, γιατί είναι θυμωμένο, γιατί βλέπετε εδώ τόσε αντιπροσωπείε, τόσε επιτροπέ που ήρθαν από τη χώρα. Τι θα μπορούσε να γίνει, δεν ξέρω. Αλλά βέβαια. πόσο έγινε μέχρι σήμερα είναι μάλλον Και εξωθείται η κατάσταση προς τη φάση του διχασμού της κοινωνίας, όπως τα είπε η Αντριάννα. σε σχέση με την ε, συνταγματική συνθήκη. Μιλήσαμε για, αυτό το, το σύνθημα του ότι ενωμένοι στην πολυμορφία, αλλά τώρα έχουμε αυτόν τον διχασμό την αντιπαράθεση βορρανότου Είναι διαλυτική η επίρρη της κατάστασης. Είδατε, στον Βασίλειο θεωρούν ότι η καλύτερη αντιμετώπιση της κρίσης είναι να φύγουν από την Ευρώπη. Άλλοι όπως στη Σκωτία τα βλέπουν αλλιώ τα πράγματα, αλλά και στην Ισπανία πολύ τώρα θεωρούν, ε, πιστεύουν το ίδιο με τους Βρετανούς. Άρα τελικά θα έπρεπε να γίνεται το αντίθετο όμως, να μας ενώνουν τα προβλήματα. Δεν θα είναι πολιτική έχουν ιστορική ευθύνη, πολύ μεγάλη σε όλη την Ευρώπη. Και από εδώ έχουν γίνει λάθη. Από αυτό το θεσμικό όργανο. Όχι, δεν είχαμε κάποιο είδους κοινωνική έκρηξη στην Ισπανία, ούτε το περιμένουμε. Αλλά κάποιοι προσπαθούν με υπόγειους, με αθέμιτους τρόπους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Ανέκαθεν συμβαίνει αυτό και στην Ισπανία και σε άλλες χώρες, ακόμα και στο Βέλγιο. Όμως, βασικός βασική μεταβλητή εδώ είναι η οικογενειακή αλληλεγγύη. Οι γονείς να βοηθούν τα παιδιά, ας πούμε, ενδιαφέρον φαινόμενο πως οι συντάξεις τώρα είναι σταθεροποιητικός παράγον. Πολλές οικογένειες τώρα τρέφονται από τη σύνταξη των παππούδων ε, μέχρι και τα εγγόνια από εκεί ζουν. Ε, γι' αυτό ακριβώ και υπάρχει αυτό το θέμα σε σχέση με το πόσο θα φυγούν οι συντάξει. Εδώ μπαίνει και το θέμα τις προεκλογικές φάσεις. Γιατί ακριβώς είναι μια κολόνα στήριξης της κοινωνίας στην Ισπανία οι συντάξει. Ήταν τρομερό πράγμα. Οι μισθοί περικόπησαν πάνω από 40% σε πολλές περιπτώσεις. Και σήμερα Πολύ. πιάνουν δουλειά με 800-900 ευρώ. Και θα πρέπει αυτοί να δώσουν εισφορά για κάποια μέρα που θα πάρουν σύνταξη που με τις, ε, με τις δημογραφικές πιέσεις και λοιπά θα πηγαίνουν στις 2.000. Είναι δηλαδή εδώ ένα παράδοξο πως όλα αυτά θα τα σηκώσει η κυβέρνηση. Γιατί όπως είπαμε, οι συντάξεις σήμερα είναι παράγον σταθεροποίησης. Είναι κατακλείδη. Υπάρχει και μια εξωτερική μεταβλητή. είναι την εντύπωση ότι η Ευρώπη και η Ισπανία κυβερνάται από τη Γερμανία. Ξεκάθαρα ανέκυψε αυτό. Και άλλωστε ποτέ δεν παρακολούθησε ο κόσμος τόσο προσεκτικά τις εξελίξεις της εκλογές στη Γερμανία όπως φέτος. είπαμε πόσο σημαντικό είναι τώρα για μας να γίνει αυτή η μεγάλη η κυβέρνηση τέλο πάντων της Εβραίου Συνασπισμού με τους σοσιαλδημοκράτες γιατί δεν είναι εντύπωση αυτό θα είναι καλύτερο για μας που χρωστάμε. Και δημιουργήθηκε τώρα πάλι η, η αίσθηση της αντιπαράθεσης βορανότου, της αντιπαράθεσης. Κακό αυτό. Αυτό πρέπει να αποφεύγεται. Πολλά πρέπει να αλλάξουν στη χώρα. Τα κόμματα θα πρέπει να, να λάβουν τις ευθύνες τους, μια που είναι θεσμοί που επικεντρώνονται περισσότερο στα ίδια συμφέροντα. υπάρχει επικοινωνία που πρέπει με τον κόσμο. Ούτε τα συνδικάτα διαδραμάτισαν το ρόλο που θα έπρεπε. Υπεραμείνονται περισσότερο των κεκτημένων, αυτών δηλαδή που έχουν δουλειά, μην τη χάσουν, παρά να κάνουν κάτι για αυτούς που έχασαν τη δουλειά τους. να προβληματιστούμε όσον αφορά το ρόλο μας, την, ε, ε, τις, ε, τι επιθυνότητα πρέπει να έχουμε τότε που ήταν τα πράγματα αλλιώ. Είχαμε όλα αυτά τα στεγαστικά δάνεια. Είχαμε αυτές τις υπερφύαλες τάσεις της αισιοδοξίας, δηλαδή τις αποφάσεις με τέτοιες συνέπειες όπως σήμερα. Επομένως θα πρέπει βαθιά να προβληματιστεί η κοινωνία. Επίσης, ο κίνδυνος στην Ισπανία τώρα θεωρώ ότι είναι αυτό το, ότι διακυβεύεται η ενότητα, ότι υπάρχει η, η ότι θα πρέπει να ισχύσει το ο σώζον εαυτόν στο θέτο. Πάντως η οικονομία πρέπει να αντιδράσει. και το ότι βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ. Δεν θα πρέπει να λέμε δόξα το Θεό και να έχουμε κάποιο είδους υπερβολική αισιοδοξία, αλλά ούτε είναι ρεαλιστική, ρεαλιστικό το να έχουμε την σημερινή άπεσιοδοξία. Ε, υπάρχουν ένα σωρό παράγοντες οι οποίοι συνυπάρχουν. Αλλά η ενότητα είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Μια που η οικονομία μας έχει τα προσόντα να ανακάμψει. Να έχουμε μια διμερούσα κοινωνία. Έχουμε την παγκοσμιοποίηση, την Κίνα, το ευρώ, πολλά πράγματα τα οποία αλλάξανε. Νομίζω ότι θα πρέπει ακριβώς τον παράγοντα ενόταν να προσέξουμε. Αυτά είχα να σας πω και ευχαριστώ να απαντήσω οποιαδήποτε τυχόν ερώτηση. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Σερβέτα. Και τώρα, θα δώσουμε το λόγο σε κάποιους από τους ετούντες. Σύμφωνα με τη μέρη σε διάταξη. Μετά τους αναφέροντες θα δώσουμε το λόγο σε βουλευτές για να και υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους προς τους εισηγητές. Πρώτα πρώτα. Έχουμε τον κύριο Θεόδωρο Τιτικάρη από την Ελλάδα αφορά το άρθρο 28 του Χάρτη Συμβουλίου των Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πιτικάρη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα, μέρα. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, ε, μέλη της Επιτροπής, ε, είδαμε ότι η κρίση ε, δεν έχει μόνο αυτά που φαίνονται, αλλά κυρίως τραντάζει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Η χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων ήταν ένας χάρτης ο οποίος ήταν προαιρετικός για τα κράτη-μέλη. Δεσμεύτηκαν μόνο ορισμένα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη που δεν ήθελαν να δεσμευθούν έκαναν opt-out στην συνθήκη τη Λισαβόνα σωματώθηκε στο πρωτογενέ δίκαιο και έγινε δίκαιο τη Ένωση, το κυρίαρχο δίκαιο. Και όμω ξαφνικά βλέπουμε ότι με παρέμβαση τη Τρόικα και μάλιστα με, το, με την στο, εφημε, δημοσιεύεται στην επίση εφημερίδα τη κυβερνήσεω στι 28 Φεβρουαρίου του 2012 καταργούνται οι συλλογικέ συμβάσει, καταργείται δηλαδή το δικαίωμα των κοινωνικών διευθυντών στον ιδιωτικό τομέα, τονίζω στον ιδιωτικό τομέα και όχι στο δημόσιο τομέα, να έχουν μεταξύ του το δικαίωμα να συνομιλούν και να συμφωνούν στο επιτρεπτό και το κατάλληλο επίπεδο αμοιβών. Ήρθε η κυβέρνηση με μια πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και κατέργησε το θεσμοθετημένο δικαίωμα των ε, σωματείων και των, οργανώσεων, ε, των εργοδοτών και των εργαζομένων να μπορούν να συμφωνούν πάνω σε ένα ουσιαστικό ζήτημα που είναι το ζήτημα των αμοιβών και το οποίο βεβαίως παίζει και σημαντικό ρόλο στο πόσο βαθιά θα είναι η κρίση. Πέρα από αυτό, ε, όπως είναι γνωστό στο άρθρο 28, πέρα από το δικαίωμα δηλαδή στις συλλογικές συμβάσεις και στις συλλογικές οργανώσεις, υπάρχει και το δικαίωμα στην απεργία. Το δικαίωμα στην απεργία στην Ελλάδα έχει καταργηθεί. Τα τελευταία χρόνια, το χρόνο του μνημονίου, έχουμε πέντε επιστρατεύσεις, martial laws, οι οποίες απαγορεύουν στους ανθρώπους να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην απεργία για να διεκδικήσουν αυτά που και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και το Σύνταγμα και ο Διεθνή Οργανισμό Εργασία έχουν θεσμοθετήσει. Τελευταία περίπτωση είναι οι καθηγητέ, είναι οι δάσκαλοι. Μάλιστα το Reuters τώρα κυκλοφόρησε με ένα τίτλο για την Ευρώπη. Ε, δεν θα τον πέραμε ποτέ να βγει ένα τίτλο για την Ευρώπη, ο οποίο έλεγε ότι η ελληνική κυβέρνηση απειλεί να βάλει του δασκάλου φυλακή αν απεργήσουν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε μια πρωτοφανή παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Βλέπουμε την ε, ε, ε, Επιτροπή που είναι ο που είναι ο θεματοφύλακας αυτών των συμβάσεων, των, των συνθέσεων που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και έχουμε φτιάξει την Ευρώπη μέχρι τώρα να διαφορεί και την Τρόικα να επιμένει ακόμα περισσότερο σε νέες περικοπές πάλι στο επιμένω στον ιδιωτικό τομέα πέρα από τα όρια και έξω από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Είμαι καλυμμένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πιτικάρη, ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Αντώνη Μπάρμπαρα Μολίνα από την Ισπανία που υπέβαλε μια ε, αναφορά για τις περικοπές ε, στον τομέα της υγείας στην Καταλωνία και στην Ισπανία γενικότερα εκ μέρους του φορέα Τεμπέους Πεσαλούτ Πούμπλικα. Καλημέρα σας κύριοι και κυρίες ε, πολίτες της ε, ε, Ευρώπης. Υποβάλαμε μία αναφορά όπου εκφράζουμε την ανησυχία μας για τις περικοπές που γίνονται στην υγεία στην Καταλωνία, λέγοντας ότι αυτή μας η ανησυχία έχει γίνει τώρα ο χειρότερος εφιάλτης. Έχουμε τόσο πολλές περικοπές αλλά οι οποίες γίνονται όλο και περισσότερο, ε, όλο και πιο σημαντικές εκθετικά και αυτό έχει επιπτώσεις και στην πολιτική υγείας στις άλλες περιοχές της Ισπανίας. Αυτές οι πολιτικές, σε αυτές τις τόσο ταραγμένες περιοχές, είναι οι ίδιες ε, πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην Καταλωνία, εφαρμόζονται παντού στην Ισπανία. Αυτή η επιδημία έχει περάσει τα σύνορά μας, είναι μια νεοφιλελεύθερη επιδημία που ε, έχουμε καταλήξει να αποκαλούμε ε, λιτοκτονία. λιτοτιτοκτονία. Η... Στην Ισπανία είχαμε ε, ένα σύστημα υγείας, αλλά η εφαρμογή αυτής, αυτού του συστήματος υγείας είχε να κάνει με τις περιοχές. Το 1993 Γι' αυτό χρειάστηκε νομοθεσία, διότι ήταν φανερό ότι αν δεν υπάρχει νομοθεσία που να εξισώνει, η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή. Αποδεχτήκαμε λοιπόν οδηγίες για τον τομέα της ε, υγείας και περιορίζεται έτσι η ισχύ των λόμπις και μειώνονται οι τάσεις ιδιωτικοποίησης οι οποίες σήμερα έχουν επανέλθει, αν και αμφισβητούνται από τους ειδικού και τις οργανώσεις. Δεν έχω χρόνο για να σας εξηγήσω τα πάντα. Δεν μπορώ να σας τα πω όλα, ένα ολόκληρο κατάλογο, αλλά θα αναφέρω επιγραμματικά αυτή τη μαύρη βίβλο των ε, σφαλμάτων και των τρομερών φαινομένων που θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε πολύ αναλυτικά. Ε, περικοπές είπαμε στον προπολογισμό, ε, λίστες αναμονής, που είναι ε, λίστες απελπισίας. Ε, κλείνουν τα χειρουργεία, οι υπηρεσίες, τα κρεβάτια, αυξάνεται η ανεργία και στον τομέα των ε, επαγγελματιών της υγείας, ασταθείς ηθικές εργασίες, επισφαλής, ε, ιδιωτικοποίησης χωρίς αναισθησία, ε, κακή φροντίδα για την υγεία των παιδιών, φτώχεια ειδικά επιστημονικά περιοδικά καταγγέλνουν την αύξηση φορέων του AIDS, ε, ε, ε, απελπισίας, κατάθλιψης, αυτοκτονιών. Από ό,τι φαίνεται θα είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση της υγείας αυτής της γενιάς από ό,τι των γονέων και παππούδων τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την υγεία και για να υπάρχει υγεία πρέπει να υπάρχει κοινωνική συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς, καλή εργασία. Ένας νέος νόμος, ένα νέο βασιλικό διάταγμα, 16-12, κάνει νέους περιορισμούς και εξαιρεί από το σύστημα υγείας πάνω από 800.000 ε, ανθρώπους που έχουν χάσει την εργασία τους, που έχουν αποκλειστεί από κοινωνία και η συμμετοχή των ασφαλισμένων αυξάνει όλο και περισσότερο για τα διάφορα φάρμακα, για φάρμακα κατά του καρκίνου, κατά των ιώσεων Αυξάνεται λοιπόν το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων. Για όλους. Δεν υπάρχει δυνατότητα να μεταφερθεί κανείς με ασθενοφόρο. Πρέπει να ε, πληρώσει κανείς για διάφορες ορθοπαιδικές ε, προθέσεις που γίνονται. Αυξάνονται οι περιπτώσεις ε, διαφθοράς, γίνονται εξεδιάντροπα αυτά τα φαινόμενα. Αυξάνονται λοιπόν οι καταθλίψεις, οι διανοητικές ασθένειες, οι αυτοκτονίες. Χρειάζεται να συνεχίσω θα, λέγατε ότι υπερβάλλω, αλλά πραγματικά δεν υπερβάλλω. Κοιτάξτε, σήμερα έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Έχουμε άρθρα επιστημονικά που επιβεβαιώνουν όλα όσα είπα. Αυτός ο δρόμος θα μας πάει απευθείας στον κρεμό, στην Άβυσσο. Η διάγνωση που κάνουμε είναι ότι η Ευρώπη είναι ασθενής. Είναι ασθενής γιατί δεν έχει την αναγκαία ψυχή του πολίτη, την αναγκαία στήριξη. Δεν κατάλαβε η Ευρώπη ότι δεν μπορεί να διαχωρίσει το βιολογικό από το ψυχολογικό και το κοινωνικό. Πρέπει να επαναδραστηριοποιήσουμε μια συνολική αντιμετώπιση της υγείας που να λαμβάνει υπόψη την ανθρώπινη διάσταση, την προσοχή, την πρόληψη, την ενημέρωση. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει επιγόντως μετάγγιση που μπορεί να γίνει μόνο μέσω της συμμετοχής των πολιτών στη δημόσια υγεία. Ως ε, ιατρός δεν μπορώ να μην σας πω ότι πρέπει και το Κοινοβούλιο να κάνει τις αναγκαίες προτάσεις για τη θεραπεία. Πρέπει να ενημερώσετε όλους όσους ενέχονται στην υγεία. Μία κοινωνία υγιής δεν μπορεί να υπάρχει αν κάποιος δεν έχει στέγη, αν δεν έχει εργασία, αν δεν έχει χρήματα για να επιζήσει. Αν δεν τα έχουμε όλα αυτά ε, τα φάρμακα δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Επιτρέψτε μου, καταλήγοντας, να πω ότι πρέπει να τα καταπολεμήσουμε όλα αυτά και να κάνω μια ερώτηση σε όλους τους ε, βουλευτές που είναι παρόντες. Αυξάνει ανισότητα. Αυξάνει η ανισότητα για τους πιο αδύναμους, τους εξαρτημένους, τους πιο ευαίσθητους. Είναι τρομερή αυτή η αδικία. Έχετε κύριοι βουλευτές συνέστηση του ιστορικού σας ρόλου που παίζεται γι' αυτό. Γιατί είναι η ε, έναρξη μιας διαδικασίας κατάργησης των δημόσιων ε, συστημάτων υγείας που καλύπτουν όλους τους πολίτες. Έχετε λοιπόν ραντεβού με την ιστορία. Γιατί να μην υπάρξει ρήτρα διαφύλαξης για την υγεία. Μια κόκκινη γραμμή που να αποτρέψει τη συνέχιση αυτής της αιμορραγίας των συστημάτων δημόσιας υγείας, τουλάχιστον όσον αφορά την ε, συνολική καθολική κάλυψη με υγιή και ισότιμο τρόπο. Καταλήγω, καταλήγω. Έλεγα λοιπόν, νονότσερε είναι, νονόκερε είναι η πρώτη υποχρέωση του ιατρού, να μην κάνει υγεία, να μην κάνει ζημιά στην υγεία. Εσείς όμως με αυτά που κάνετε, κάνετε ζημιά στην υγεία. Πρέπει να υπερασπιστούμε τη δημόσια υγεία, πρέπει με βάση την ιστορία και την επιστήμη να καταλάβουμε ότι είναι η ουσιαστικότερη υπηρεσία, η ουσιαστικότερη συμβολή στην ανάπτυξη της κοινωνίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ κύριε Μολίνα. Περνάμε στην τρίτη αναφορά. Η κυρία Σάρο Καμπονοκάσας, η οποία θα μας παρουσιάσει την αναφορά για τις καταχρήσεις που έγιναν από ένα ταμιευτήριο της Ισπανίας με έξι καταγγέλλοντες. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα σας εξηγήσω περί τίνος πρόκειται από το λεξικό της Real Academia τι σημαίνει απάτη. Είναι μια, ένα γεγονός το οποίο οδηγεί σε ζημιά και γι' αυτό ακριβώς τον Απρίλιο που μας πέρασε απευθύνθηκα σε εσά στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο πατέρας μου είναι θύμα, όπως και πολλοί άλλοι Ισπανοί πολίτες, της απάτης που έγινε με την ε, πώληση προνομιούχων μετοχών όπως λέγονται, που πουλήθηκαν σε μικρούς αποταμιευτές από μια Ισπανική τράπεζα που ακούει στο όνομα Μπάνκια. Πριν ε, από 1,5 χρόνο ο πατέρας μου και όλοι οι υπόλοιποι αγωνίστηκαν για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους, δηλαδή τις αποταμιεύσεις τους που νόμιζαν ότι ήταν εγκυμένες. Δυστυχώς όμως δεν ήταν. Και στάλει μία επιστολή από το κράτος που εξηγούσε την καταγγελία και έφτασε βέβαια στην τοπική εισαγγελία της Βαρκελόνης, η οποία όμως δεν μας έχει στείλει καμία απάντηση. Ρωτάμε λοιπόν, Πρόκειται για διαφορία, πρόκειται απλώς για παθητική στάση και μετά τελίτσες, τελίτσες, τελίτσες. Επίσης ήρθαμε σε επαφή μαζί σας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί έχουμε την αίσθηση ότι οι επίσημοι οργανισμοί του Ισπανικού κράτους, οι θεσμοί δηλαδή στην Ισπανία, διαφορούν για μας, δεν μας στηρίζουν. Ήρθαμε σε επαφή με δικηγόρους, με οργανώσεις καταναλωτών και σχετικά με αυτή την πρόταση της Βάνκια και Διατησία. Ο πατέρας μου λοιπόν ζήτησε τη διαιτησία αυτή τον Ιούλιο που μας πέρασε. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει γίνει καμία διαιτησία. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε βεβαιότητα. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να λυθεί θετικά το θέμα αυτό, η διαιτησία. Αλλιώς θα πρέπει να πάμε στα δικαστήρια με ό,τι αυτό σημαίνει. Θα ήθελα να υποστηρίξετε περισσότερο τα δικαιώματά μας εμάς των πολιτών και των καταναλωτών για να μην επαναληφθούν τέτοιες καταστάσεις, να νιώθουν οι πολίτες δηλαδή ότι έχουν εξαπατηθεί από την τράπεζα στην οποία έχουν εμπιστευθεί τις αποταμιεύσεις μια ολόκληρης ζωής, τα χρήματα τα οποία τόσο τίμια κέρδισαν. Ερωτήσεις έχουμε πολλές. Η κυβέρνηση τι κάνει, ποιοι είναι υπεύθυνοι για την απάτη αυτή, γιατί δεν τους πάνε στα δικαστήρια, γιατί επιτράπηκε να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση κλπ. κλπ. Πώς θέλουν τα, οι πολίτες να πιστεύουν στην κυβέρνηση όταν μας απογοητεύουν οι κυβερνήσεις τόσο. Εμείς θέλουμε οι υπεύθυνοι για την απάτη αυτή να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να υπάρξει δικαιοσύνη, να τηρηθεί ο νόμος. Και κυρίως επειδή η απάτη αυτή έλαβε χώρα μέσα στην καρδιά της κρίσης. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Καμπουθάνο. Τώρα, τρεις, ο κύριος Σάλβας, Τσουκαλάς και ο κύριος Σαλαβράκος έχουν ζητήσει το λόγο και ο κύριος Γιάρ και εγώ θέλω να παρέμβω παρακαλώ. Ο κύριος Πάλος Σάλβα πρώτα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θέλω να αναφερθώ στην κυρία Καπουθάνο αυτά που είπε πριν από μερικές εβδομάδες, μήνες, ενημερώθηκα. Πρώτα απ' όλα θέλω να τη εκφράσω κάθε συμπαράσταση και συμπάθεια για αυτά τα οποία αναφέρει για τον πατέρα της. Πράγματι υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Το θέμα των προνομιούχων μετοχών πρέπει να ξέρουμε ότι είναι μια πραγματική τραγωδία καρπός μιας ελαστικής νομοθεσίας της κυβέρνησης, της προηγούμενης που δημιούργησε το πρόβλημα και η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί, αντί να κρύβεται, προσπαθεί να βρει λύση αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα. Τώρα τι λύση. Όπως ακούσαμε, τις περισσότερες φορές η λύση βρίσκεται με διαιτησία. Κάτι το οποίο εφαρμόζει ο σύστημα πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση της Γαλήθια. Από εκεί ξεκίνησε η λύση αυτή μέσω διαιτησίας. Θέλω επίσης να σας πω ότι προσπαθώντας να πετύχει λύσεις και η κεντρική κυβέρνηση αλλά και οι περιφερειακές κυβερνήσεις να ξέρετε ότι έχει περιορισμούς. Την περιορίζει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Επίτροπος Αρμόδιος για, την, για τον ανταγωνισμό, ο κ. Σαλμούνια. Τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι αν η κυβέρνηση αποφάσιζε αύριο, ας πούμε, ότι όλοι όσοι πιστεύουν ότι πρέπει να ληφθεί μια απόφαση και η κυβέρνηση πει εντάξει θα επιστρέψει τα χρήματα, να επιστρέψουν τα χρήματα, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα συμφωνήσει. Οπότε επιμένω για το ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει λύσεις, οι οποίες όμως λύσεις θα είναι έτσι κι αλλιώς υπό προϋποθέσεις τις οποίες βάζει ο αρμόδιος Επίτροπος Ανταγωνισμού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο διευθυντής τώρα ο Αντώνιο Καρασκόσα είπε ότι 70% περίπου όσων έχουν τέτοιες προνομιούχες μετοχές στα χέρια τους θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Συνεπώς, επιμένω ότι το πρόβλημα βρίσκεται προς τη λύση του, πάει προς τη λύση του. Η κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να βρει λύση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως πολλές φορές εκφράζει αμφιβολίες για το κατά πόσο κάποιοι από τους επενδυτές, από αυτούς που είχαν προνομιστικές μετοχές και είχαν την ενημέρωση, μπορεί να επωφεληθούν από τη διατησία. Είναι ένα πρόβλημα που πάντως προσπαθούμε να το λύσουμε και η κυβέρνηση αλλά και διάφορες αυτόνομες κυβερνήσεις στην Ισπανία θα προσπαθήσουν να το λύσουν το ζήτημα. Επιμένω για άλλη μια φορά ότι έχει την πλήρη αλληλεγγύη μου η αναφέρουσα, η οικογένειά της, ο πατέρας της και θέλω να την καθησυχάσω γιατί το πρόβλημα αυτό θα λυθεί κυρίως για όλους εκείνους τους επενδυτές οι οποίοι καλή την πίστη έδρασαν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τσουκαλάς παρακαλώ. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους διακεκριμένους ομιλητές μας, αλλά επίσης τους ετούντες, οι οποίοι περιγράφουν ένα τοπίο που λίγο πολύ φαίνεται να έχει τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά σε όλες τις χώρες του Νότου της Ευρώπης με ακραία περίπτωση τη χώρα μου, δηλαδή την Ελλάδα. Θα ήθελα να κάνω δύο-τρεις παρατηρήσεις. Πρώτη παρατήρηση η κυρία, η ερήτημος Ιταλής κυρία αναφέρθηκε στο μαγείρεμα των στατιστικών στοιχείων της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με τα δημοσιονομικά της. Σοβαρά αμφιβάλλω αν η ανίκανη ελληνική δημόσια διοίκηση ή το απαξιωμένο πολιτικό κατεστημένο θα μπορούσε χωρίς τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδεχθεί τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και τα οποία πολύ αργότερα φάνηκε να είναι απατηλά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία ρήξη ανάμεσα σε βορρά-νότο. Η ρήξη, η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε βορρά-νότο είναι πολύ πιο μόνιμη από ό,τι φαίνεται. Και δεν, γιατί δεν πρόκειται για οικονομική ρήξη. Πρόκειται για τεχνολογική ρήξη πρόκειται για διαφορά ανάπτυξης. Για να αποδείξω αυτό που λέω, αν πάρετε την Ευρώπη των 28 και αν πάρετε την Ευρώπη των 7 υγιών οικονομιών της Ευρώπης, θα δείτε ότι η μεν Ευρώπη των 28 υστερεί τεχνολογικά σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν έχει πρωτιά, ενώ οι 7 υγιείς οικονομίες με μεγάλη βιομηχανική και τεχνολογική παράδοση, δηλαδή Σουηδία, Φιλανδία, Γερμανία, Ολλανδία και ούτω καθεξής, αποτελούν πρωτοπορία παγκοσμίω. Πρέπει να καταρρέψουμε και ένα μύθο, τον μύθο ότι χρηματοδοτούν οι βόρειοι τις οφειλές των νοτίων. Εγώ έχω υπόψη μου τουλάχιστον δύο επώνυμες δηλώσεις Υπουργών Οικονομικών τόσο της Γερμανίας όσο και της Αυστρίας που διαβεβαιώνουν τους πολίτες τους ότι από αυτήν την κρίση οι πολίτες κερδίζουν και μάλιστα αν θυμάμαι καλά είχαν δώσει και ε, τα ποσά τα οποία κέρδισε η Γερμανία και η Αυστρία από αυτήν την κρίση. Τέλος, ανέφερε ο γιατρός από την Ισπανία, τον οποίον ευχαριστώ θερμά για την εισήγησή του, σχετικά καθώς επίσης και ο Ισπανός δημοσιογράφος, σχετικά με το ζήτημα των συντάξεων ως παράγοντα σταθεροποίησης. Στην Ελλάδα τα ασφαλιστικά ταμεία κουρεύτηκαν με αποτέλεσμα αυτός ο σταθεροποιητικός παράγον να είναι αμφίβολο αν θα υπάρξει, αν δηλαδή τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας μου θα μπορούν να πληρώσουν συντάξεις που κατά τη δήλωση των εισηγητών αποτελούν σταθεροποιητικό παράγοντα. Τέλος, πρέπει να σας αναφέρω ότι δεν έχω τις ειδικέ γνώσεις να μπορέσω να δώσω μια πλήρη περιγραφή της κρίσεως ως θετικός επιστήμον εξακολουθώ να διαμαρτύρομαι όποτε οι αριθμοί έχουν προήγηση έναντι των ανθρώπων και όποτε τα μοντέλα επιβάλλονται στην πραγματικότητα. Αυτό είναι αντίθετο στη φυσική αιτιότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει. Επομένως, μην εκπλήτεστε ότι ξαφνικά στην Ήπια και μιλήχια Ελλάδα ξεφυτρώνουν παραστρατιωτικές οργανώσεις της χιδεότητας της χρυσή αυγή και σας παρακαλώ να θυμηθείτε ότι σε καιρούς δυσκολίες σε άλλες χώρες της Ευρώπης τέτοια χαρακτηριστικά τα είχαμε επίσης. Δεν θέλω να αναφέρω επωνύμως, αλλά μη μου πείτε ότι δεν θυμάστε παραστρατιωτικές νεοναζιστικές οργανώσεις σε χώρες που τώρα κάνουν τον κίνσορα της δημοκρατίας και ας μην ξεχνάμε ότι μια τέτοια, ένα τέτοιο πολιτικό μόρφωμα κυβερνάει σε μια βόρεια χώρα της Ευρώπης. Θέλω να κάνω μια έκκληση. Φαίνεται στην Ευρώπη αυτό τον καιρό να γίνεται με λεφτά ό,τι γίνει και στην Αμερική με αίμα. Εάν πρόκειται να επαληθευθούν αυτά που οι συνάδελφοι είπαν στον κύριο Μπαρόζο, πως δηλαδή μέσα σε μία θητεία από 74% των πολιτών που ήταν υπέρ της Ευρώπης, 74% ανακαλύπτουν ότι η Ευρώπη αποτελεί το πρόβλημα, θα έχουμε την αποτυχία του πιο φιλόδοξου ανθρώπινου πειράματος, του πειράματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή το μαλαντέτο φιόρε του Δάντι έχει κάνει να είναι όλη η Ευρώπη Σέρβα και όχι μόνο η Ιταλία ή η Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσουκαλά. Να συνεχίσουμε με τους άλλους συναδέλφους. Ο κύριος Αλαβράκος. Πρόεδρε, ε, άκουσα με προσοχή όλους τους ομιλητές ε, και πάνω από το βήμα και κάτω από το βήμα. Και συμφωνώ περίπου σε όλα τα οποία ανέφερα. Θέλω να επενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε με το ρομαντισμό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τον ενθουσιασμό και την αισιοδοξία για να κάνουμε μια Ευρώπη καλύτερη για τους Ευρωπαίους, μια ενωμένη Γερμανία εδώ και 20 χρόνια που την βοηθήσαμε πάρα πολύ όλοι και φτάσαμε στο σημείο του ρεαλισμού του σημερινού που δεν μπορούμε να τον διαχειριστούμε. Διότι απεδείχθη ότι αυτή τη στιγμή ήρθε κρίση στην Ευρώπη, η διαχείριση αυτή της κρίσεως διέσπασε και τις δομές αλληλεγγύης αλλά παράλληλα και την εμπιστοσύνη του ενός προς τον άλλον από τα κράτη-μέλη. Τώρα έχει φτάσει και στους πολίτες. Και συμφωνώ μαζί σας ότι αν κάτι είναι αναγκαίο για την Ευρώπη, για την Ευρώπη του μέλλοντος, είναι η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη χωρίς ο ένας όμως να είναι βάρος στον άλλον. Χωρίς το ένα κράτος μέλος να είναι βάρος σε ένα άλλο κράτο μέλος. Όμως από όλη την κουβέντα ε, δεν είδα προτάσεις. Τα διαπιστώσαμε όλα αυτά τα πράγματα. Και στις διαπιστώσεις μας έλειψε ένα κεφάλαιο που είναι η δημογραφία που έχει μεγάλη σημασία διότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη αποτελεί το 8% του παγκόσμιου πληθυσμού και περίπου το 30% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Το 2035 όμως η Ευρώπη θα είναι περίπου το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού, ίσως και λιγότερο, και υπολογίζεται το ΑΕΠ της Ευρώπης να είναι στο παγκόσμιο ΕΠ περίπου το 15 έως 18%. Δηλαδή η Ευρώπη φτωχαίνει. Και επομένως πρέπει πρώτον να διατηρήσει τη συνοχή της διότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις νέες εξελίξεις από τα αναδυόμενα κράτη και το δεύτερο πρέπει να αυξήσει το ευρωπαϊκό εισόδημα προ την κατεύθυνση τη αυξήσεω του ευρωπαϊκού εισοδήματο, εγώ τα τελευταία πέντε χρόνια δεν βλέπω τίποτα. Το να διατηρήσουμε αυτά τα οποία έχουμε πρέπει να κάνουμε προσπάθειες να τα διατηρήσουμε. Αλλά για να τα διατηρήσουμε πρέπει να αυξήσουμε το εισόδημα και προς αυτή την κατεύθυνση δεν βλέπω τίποτα. Και θα σας παρακαλούσα σαν κοινωνική φορείς να επανέλθετε με προτάσεις του τι πρέπει να κάνουμε στην Ευρώπη. Πρόχειρα εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκω ότι το 25%, τα 25 εκατομμύρια ανέργων στην Ευρώπη δεν μπορούμε να τα απορροφήσουμε. Μιλάμε για καλυτερέψη της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών με 25 εκατομμύρια ανέργους, Ευρωπαίους ανέργους, ε, γιατί υπάρχουν και οι παράλληλοι άνεργοι ε, οι οποίοι προέρχονται από έμικρος ε, και προς αυτή την κατεύθυνση δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να ανοίγουμε ούτε τις μισθές της εργασίας. Μήπως θα πρέπει να προσανατολιστούμε σε μια πανευρωπαϊκή πολιτική που να έχει επιστροφή σε στοχευμένο, σε στοχευμένο πάντα λέω, πρωτογενή τομέα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε πληθυσμούς και σε θέσεις εργασίας και σε παραγωγική εργασία και σε χρήσιμη εργασία δι' ενόψη του γεγονότος ότι ε, οι τάσει είναι τα τρόφιμα κυρίως παγκοσμίω να αυξάνουν. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να το δούμε το πράγμα πιο ρεαλιστικά. Ε, στο συναισθηματικό τομέα όλοι συμφωνούμε αλλά να διακυβερνηθεί ένας τόπος ή ένας χώρος χρειάζεται ρεαλισμός. Και θα κλείσω με το εξής τελευταίο. Ε, συνήθως ε, οι άνθρωποι, πολλές φορές τα κράτη, πολλές φορές και οι ιδεολογίες, έχουν την καλύτερη άποψη για τους εαυτούς τους. Παράλληλα όμως έχουν και τη χειρότερη άποψη για τους άλλους. Αυτό είναι το λάθος. Αυτό είναι η επιρρεπής ασθένεια των βλακών να μην γίνουμε βλάκες, να μην μείνουμε βλάκες και να μην είμαστε όλοι ε, στις θέσεις τις οποίες έχουμε και να μην κάνουμε κανένα βήμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σαλαβράκο. Να υπενθυμίσω σε όλους ότι έχουμε άλλο δύο τμήματα της συζήτησης. Παρακαλώ οι παρεμβάσεις να είναι προσαρμοσμένες στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Ο κύριος Πέτερ Γιάνν παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ε, υποβάλλοντας αναφορές. Καλό είναι που έχουμε δυνατότητα να το συζητήσουμε για να βρούμε θετικές ε, διατυπώσεις. Είμαι πολιτικός και πρέπει να εξετάζω τα πράγματα όσα έχουν. Βεβαίως προσπαθούμε να δούμε τις θετικές πλευρές της κατάστασης. Ας ξεκινήσω λοιπόν ε, με τα θετικά. Η κρίση την οποία ανηφιστάμεθα είναι η πραγματική δοκιμασία για το εάν μπορούμε να επιζήσουμε. Γιατί είχαμε, είχαμε υποσχεθεί ε, οι μεν στους δε ότι και στους καλούς και στους κακούς καιρούς θα στηρίξουμε τον, ο ένας τον άλλον. Τώρα που δεν είναι καλή η καιρή θα πρέπει να δούμε αν έχουμε την εσωτερική δύναμη να υπερβούμε την κρίση. Το πρόβλημα ή μάλλον τα δύο προβλήματα και σε σχέση με την πρώτη ε, εισηγήτρια. Πώς να το πω. Πρέπει κάποια στιγμή να αναγνωρίσουμε και τα δικά μας λάθη. Αυτό που δεν ε, άκουσα από κανένα ήταν ε, να πούμε ποια είναι η δική μας ευθύνη. Γιατί δεν είναι θεομηνία αυτό που μας συνέβη. Υπάρχει μια προϊστορία. Έκαναν κάποιες κυβερνήσεις κάποια λάθη. Πρέπει να τα παραδεχθούν. Τι λάθη έκαναν. Εάν δεν το κάνει κανείς αυτό, καταλαβαίνω βεβαίως ε, αυτούς που έχουν ε, αυτή την εντύπωση ότι ε, κάποιοι έβγαλαν λεφτά και κάποιοι τώρα πρέπει να πληρώσουν τα σπασμένα. Τώρα βέβαια ισχύει αυτή η εντύπωση έχει τη σημασία του, αλλά αν δεν υπερβούμε αυτή τη φάση δεν θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να κάνω έκκληση προς όλους, πρέπει να το συζητήσουμε μεταξύ μας, να κάνουμε διάλογο. Βεβαίως να υποστηρίξουμε τους αδύνατους, είμαστε Επιτροπή Αναφορών. Βεβαίως ε, και τις τράπεζες πρέπει να βοηθήσουμε. Είδαμε τι έγινε με την ε, Lehman Brothers. Όταν ε, πτώχευσε η Λίμαν, οι Γερμανοί είπαν ε, «Α, καλά, είναι Αμερικανική τράπεζα, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά διαπιστώσαμε πως είναι παγκόσμιο πρόβλημα». Αλλά δεν είναι αυτός σκοπός η βοήθεια στις τράπεζες. Ε, τις βοηθάμε τις τράπεζες για να βοηθήσουν τους μικροεπενδυτές, τους μικροκαταθέτες. Να τους δώσουμε εγγυήσεις και βεβαίως και για τα ακίνητα να διατηρήσουμε την ιδιοκτησία των μικροϊδιοκτητών. Αυτό που δεν επιτύχαμε και ίσως ε, να υπάρξουν προτάσεις ε, για τα θέματα αυτά από τους συζητητές είναι να περιγράψουμε την ε, αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη έχει δύο πλευρές. Από τη μία δίδεται βοήθεια, αυτονόητο, πρέπει να βοηθήσουμε ορισμένα άτομα, ορισμένες πλευρές, αλλά πρέπει να υπάρξει και αυτοβοήθεια. Δηλαδή βοηθάμε κάποιους, αλλά και αυτοί να βοηθούν τον εαυτό τους. Αλλά εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν υπήρξε επαρκής επικοινωνία. Αυτοί που βοηθάνε έχουν την εντύπωση ότι κάνουν ό,τι μπορούν, κάνουν παραπάνω από ό,τι μπορούν, αλλά εκείνοι που λαμβάνουν τη βοήθεια θεωρούν ότι λαμβάνουν ε, ανεπαρκή βοήθεια και ότι όλα αυτά πάνε στράφη. Αναφέρθηκε το λεγόμενο σχέδιο Marshall, υπόθηκε ότι είναι εντελώς λάθος πολιτική που ακολουθούμε, από ευρωπαϊκή πλευρά και ως βουλευτής από τη Γερμανία από ένα συγκεκριμένο ομόσπονδο κράτος ξέρω ότι δεν αρκούν οι χρηματοδοτήσεις για να ανορθωθεί η οικοδομία. Οπότε, βεβαίως, καλές οι επενδύσεις, καλό το σχέδιο Μάσον, καλή η ε, ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά χρειαζόμαστε συγκεκριμένα προγράμματα. Γιατί ξέρετε, χρήματα υπάρχουν. Ε, ε, δεν ισχύει ότι δεν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Είπαμε, η Ευρώπη θέλει να βοηθήσει την ε, καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, αλλά πρέπει να γίνει με συγκεκριμένο τρόπο αυτό. Κοιτάξτε, εδώ είναι τα χρήματα, πού είναι τα προγραμματά σας, πώς θα τα δαπανίσουμε, θα τα αξιοποιήσουμε αυτά τα χρήματα. Αυτά πρέπει να έχουμε. Βεβαίω, αυτό θα βοηθήσει να υπάρξει αίσθημα αλληλεγγύης και να υπάρξουν και επαρκείς επενδύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πίτερ. υπενθύμησα και προηγουμένως ότι έχουμε άλλο δύο, άλλα δύο τμήματα της συζήτησης και θα έχει δυνατότητα να ξαναλάβεις το λόγο αν χρειαστεί. Μάργαρετ, παρακαλώ έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι με προκάλεσαν. Με προκάλεσε βασικά η πρώτη ομιλία που άκουσα που αναφέρθηκε η ομιλήτρια στο ρήγμα ανάμεσα στο Βορρά και τον Νότο, που είπε ότι ο Βορρά είναι που τιμωρεί, που κυριαρχεί, που κάνουν τους καθολικούς τον Νότο να υποφέρουν. Εγώ έρχομαι από τη Δανία, από το Βορρά, λοιπόν. Ε, τουλάχιστον από το Βορρά, στον οποίο αναφέρθηκε η ομιλήτρια ή μάλιστα ακόμα και πιο βόρεια. Εν πάση περιπτώσει, όχι, δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε. Δεν έχουμε αυτές τις ιδέες για τιμωρία. Όχι, έχουμε άλλες ιδέες. Εγώ πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι στις βόρειες χώρες πιστεύουν ότι οι ισχυρές οικονομίες επωφελήθηκαν από το σταθερό νόμισμα. Από το γεγονός ότι δεν μπορείς να υποτιμήσεις το νόμισμά σου. Δεν είναι κάτι καινούριο. Το ξέρουμε αυτό. Αυτό όμω που χρειαζόμαστε είναι πιο επικοδομητική κριτική. Κριτική και απέναντι στις βόρειες χώρες, τόσο τη δικιά μου όσο και τη Γερμανία. Γιατί προφανώς υπήρξε έλλειψη οράματος και ενωτόμου στρατηγικής για επενδύσεις. Στην καλύτερη των περιπτώσεων αυτό που έγινε είναι ότι οι άνθρωποι επειδή εκεί έχουν τα καλύτερα λόμπι κοίταξαν τις παλιές παραδοσιακές βιομηχανίες, τους παραδοσιακούς κλάδους. Δεν ακολουθήσαμε στρατηγικές επενδυτικές για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν υπήρξε για μένα ε, κακό όραμα. Μόνο αποταμιεύσεις σκεφτόμαστε ή τις παλιές παραδοσιακές βιομηχανίες. Τώρα με τις γερμανικές εκλογές όλοι ελπίζουμε ότι η Γερμανία θα αλλάξει κάπως αυτήν την στρατηγική. Αν μη τι άλλο, στη Δανία, αυτό είναι το πρώτο που έχουμε στη δικιά μας σε διάταξη. Οπότε εμείς δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε τις νότιες χώρες. Εγώ έχω συνεργαστεί πολύ με Ισπανούς και με την Ισπανία. Εντάξει, υπάρχει διαφθορά. Είναι δύσκολο να ακούς κάποιον να μιλάει για διαφορές στην οτροπία και να αναφέρεται στη διαφθορά. Μα η διαφθορά δεν είναι οτροπία, είναι αδίκημα και πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν τέτοιο. Επιμένουμε λοιπόν στη διαφάνεια όλων των θεσμικών οργάνων. Φορολογία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσουμε τους δικούς μας φορολογούμενους να πληρώνουν για κάποιον ο οποίος δεν εξηγεί τι έγιναν τα χρήματα τα οποία είχε. Παράδειγμα, Ιταλία. Η Ιταλική κυβέρνηση είναι βέβαια μια διαφορετική ιστορία. Εγώ κοίταξα και στο παρασκήνιο και τελικά υπάρχει μεγάλη ανευθυνότητα στην Ιταλική δίκηση. Το γεγονός ότι στην καμπάνια ένας περιφερειακός υπουργός χρειάζεται συμφωνία από 561 δημάρχους για να κάνει κάτι, ε, πώς να γίνει αυτό το κάτι. Είναι αδύνατον. Άντε δεν να πολεμήσεις και με τη μαφία. Στη ΔΕΝ Ελλάδα δεν έχουμε φορολογικό σύστημα. Δεν είναι ότι θέλουμε να τιμωρήσουμε τους Έλληνες και γι' αυτό επιμένουμε να έχουν φορολογικό σύστημα. Όχι. Είναι γιατί χρειάζονται. Και γιατί έτσι προσπαθώ και εγώ να πείσω τους δικούς μου πολίτες να πληρώσουν για το δημόσιο χρέος. Σας φαίνεται ανόητο αυτό. Στην Νότια Ευρώπη με την αποκέντρωση κοντά στον πολίτη καταλήγουμε σε διαφθορά. Μπορεί να μην λέγεται μαφία, αλλά υπάρχει διαφθορά. Αν συνεχίσετε σε αυτή τη γραμμή δεν πρόκειται πράγματι να καταλήξουμε πουθενά. Υπάρχουν κάποια όρια. Εγώ αντιλαμβάνομαι τα όρια της Βόρειας Ευρώπης Μπορεί να κατηγορώ την Βόρεια Ευρώπη για πολλά πράγματα, αλλά έχω πολλά να πω και για την Νότια Ευρώπη. Κάτι λοιπόν πρέπει να γίνει για να διορθωθούν τα συστήματα τα οποία δεν λειτουργούν καλά. Ξέρω Δανούς οι οποίοι ζουν στην Ισπανία 10-30 χρόνια, όχι από τη δικιά μου πολιτική οικογένεια, και μου λένε γιατί να πληρώσει κανείς φόρους αφού δεν έχει σημασία τελικά. Ε, αυτή την ε, γλώσσα ή την οτροπία αν θέλετε να την αλλάξουμε. Αν και εμένα δεν μου αρέσει να την ονομάζουμε νοτροπία αυτή τη στάση. Ο Πρόεδρος, κύριε Άκη, ευχαριστούμε. Κύριε Μπριστάνο, το λόγο παρακαλώ να είστε σύντομος, διότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και να δώσουμε το λόγο στους άλλους αναφέροντες, ε, στους ε, εισήγητες του πάνελ και σε όλους. Μπού στην άρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα συστήσω εδώ τη σύγκρουση των ε, ε, εθνών και των πολιτισμών, γιατί ε, αν το κάνουμε αυτό, τότε δεν βγαίνουμε πουθενά. Πάει η Ευρώπη, εάν αυτό έχει ως αφετηρία τη σύγκρουση. Δεν κάνουμε τίποτα έτσι, αλλά αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, είναι Ποια είναι η επίπτωση, ποιε είναι οι συνέπειε τη κρίση για την Ευρώπη και για του Ευρωπαίου. Πρόκειται για μια διαδικασία που μεγαλώνει τι ανισότητε μεταξύ των κρατών μελών και μέσα σε κάθε κράτο μέλο. Στον παλιών και των νέων κρατών μελών το μόνο που γίνεται είναι να αυξάνει η απόσταση, η ανισότητα. Άρα αυτό πάει να πει ότι η πολιτική της συνοχής δεν φέρνει ως συνέπεια αυτά τα οποία έπρεπε λόγω αυτή της αιμονίας στη λιτότητα. Δεύτερον. Και μεταξύ των κοινωνικών ομάδων μου λένε και περισσότερε ανισότητε, γιατί ποτέ μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν είχαμε τέτοιε ανισότητε μεταξύ των Ευρωπαίων. όλο ένα και περισσότερο με κάποιους πάρα πολύ πλούσιους και όλο ένα και περισσότερους που είναι και κάποια από την ε, μεσαία τάξη. Γιατί εξαθλίωσε δηλαδή της μεσαία τάξης. Κάτι το οποίο ποτέ δεν έχει ξανασυμβεί. Ένα τρίτο στοιχείο. μια εντυπωσιακή μείωση της δυνατότητα πρόσβασης ε, των Ευρωπαίων στην παιδεία και στις υπηρεσίες ε, υγείας. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τη δική μου χώρα, τη Ρουμανία. Και σε άλλες χώρες ισχύει το ίδιο. Αποστέρηση δηλαδή των Ευρωπαίων από τα βασικά του δικαιώματα που είναι το δικαίωμα στην παιδεία και στην δημόσια υγεία. Εάν συνεχιστεί έτσι, τότε έχουμε τώρα την πιο σημαντική επίπτωση που αφορά την πολιτική. Οι πολιτικές ελίτ έχουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο το ότι τώρα δεν υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη του κόσμου προς ε, του, τους θεσμούς και προς τα κόμματα, αλλά όλο ένα και περισσότερο αναδύονται και αποκτούν περισσότερο κύριο σε διάφορε ακραίε ομάδε, αρχικές ομάδε. Λάβετε υπόψη τι συμβαίνει στην ε, Ελλάδα αλλά και πολλέ φορέ και στη Γερμανία που έχουμε αυτέ τι ριζοσπαστικέ, τι ναζιστικέ ομάδε. Μα και στη δική μου χώρα. Ε, το βασικό πρόβλημα είναι το ότι έχουμε εντυπωσιακή συρρήκνωση της ε, εμπιστοσύνης του κόσμου προς τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα, προς τους θεσμούς που αυτά ήσαν οι πρωτοπόροι που οικοδόμησαν την Ευρώπη. Άρα τελικά το ερώτημα είναι πώς κανείς θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Του χρόνου έχουμε εκλογέ. Εκεί θα έχουμε κατά κάποιο τρόπο την ακτινογραφία της ευρωπαϊκής κοινωνίας και το κάθε κοινοβούλιο που ήταν ε, η Ακρόπολη, το ήταν το, το, το κάστρο της αντίστασης κατά της φιλοσοφίας της λιτότητας. Εάν λοιπόν το, αυτό το κοινοβούλιο εδώ πέρα γίνει πιο προβληματικό, γίνει λιγότερο φιλοευρωπαϊκό, τότε όλο το ευρωπαϊκό όραμα της εν κινδύνο. Άρα θα πρέπει όλους αυτούς τους πράγματες να τους λάβουμε υπόψη. Όλους μαζί. Σε ένα τοπίο το οποίο είναι πάρα πολύ απειλητικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το ευρωπαϊκό όραμα. Τι είπε ο Μαλουρό, ξέρετε είτε θα έχουμε κοινωνική Ευρώπη και έτσι να μπορούν οι Ευρωπαίοι να έχουν εμπιστοσύνη, να μπορούν να ποντάρουν στο ευρωπαϊκό όραμα. αλλιώ τότε θα ε, εξαλωθεί, θα, θα γκρεμιστεί το ευρωπαϊκό όραμα. Ευχαριστούμε κύριε Κωστινάρου. Τώρα να δώσουμε το λόγο στους αναφέροντες, αλλά πρώτα στα μέλη του πάνελ. και θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι είχαμε πει πριν από ένα χρόνο γιατί ότι μπορεί να πτωχεύσουν κάποιες χώρες να έχουν το ευρώ και τίποτα δεν έγινε από αυτά γιατί πέρσι ε, είχαμε όλες αυτές τις ε, αναταραχές, τα φυτέψαμε πίσω μας και οι αλλαγέ τώρα στι χρηματοοικονομικέ αγορέ ε, έχουν επιπτώσει την πραγματική οικονομία. Γιατί σα τα λέω όλα αυτά, Γιατί η πολιτική λέμε πολλά, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να προτείνουμε και κάποιε λύσει. Οπότε, μεταξύ των μέσων πρέπει να πάρουμε με βαθμίο τρόπο είναι το πώ θα έχουμε κάποια βιωσιμότητα των δημοσιονομικών σε όλα τα κρατημέλη. Να έχουμε κάποιε μεταρρυθμίσει που θα πρέπει να γίνουν σε διάφορα κρατημέλη τη Ένωση εκεί που διαπιστώνεται ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. από αυτή την ε, αποσταθεροποίηση εκείνων των χωρών όπως διαπιστώνουμε. Να, και στη χώρα μου. Όπως ε, γνωρίζουμε πως πολλοί είπαν για το τι γίνεται στην Ισπανία. Ας μην ξεχνάμε ότι όταν ανέβηκε στην εξουσία αυτή η κυβέρνηση το 2012 αντιμετώπιζε μια κατάσταση τραγική και προσπάθησε να συγκρατήσει την κατάσταση στα δημοσιοοικονομικά, σκληρά μέτρα, φέραν θυσίες πολλές για τον Ισπανικό λαό. Όμως ε, οδήγησαν στο να σωθεί η Ισπανία, ε, είχαμε κάποια, κάποια συγκράτηση του ελλείμματος είχαμε την αναδιάρθρωση του δημοτοοικονομικού μοντέλου στην Ισπανία, που τώρα είναι τόσο χρόνια και επίσης είχαμε την πιο φιλόδοξη αλλαγή και τις μεταρρυθμίσεις και τα αποτελέσματα τώρα είναι ξεκάθαρα. Είχαμε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αυτό φαίνεται στο, στους διάφορους κλάδους της οικονομίας. Είδαμε τη γίνεται στους ισοζυγείο πληρωμών που για πρώτη φορά φτάσαμε σε πλεόνασμα από το 97 και το έλεγε ο κ. Σαλαβράκος το τι μέτρα πρέπει να πάρει κανείς. Να, κάποια από αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν προταθεί και τώρα δώσουν πάνω σε αυτό το λόγο στους ε, αγρότες του πάνελ. Επίσης θέλω να πω για την κυρία Άουκιν σε σχέση με αυτά τα οποία μας είπε στον αφορά την Ισπανία. Ξέρω ότι αγαπάει τη χώρα μου η κυρία Άουκιν. Της αρέσει να ασχολείται με την Ισπανία, αλλά μην ξεχνάτε κυρία Άουκιν, αγαπητή φίλη Μάργαρετ, ότι όλα υπάρχουν παντού. Δηλαδή ότι υπάρχουν όντως κάποιοι παράλογοι νόμοι, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που είναι πάρα πολύ λογικοί και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όμως και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και στην Ευρώπη ισχύουν για όλο τον κόσμο και πάρα, πολλά προβλήματα που συζητούμε στην Επιτροπή των Αναφορών προέρχονται από τη δική σας χώρα, τη Δανία. Δεν βγαίνει πουθενά να τον αρχίσουμε τη ζήτηση αυτή τη βάση. Οπότε, να δώσουμε το λόγο τώρα στους τρεις αναφέροντες να είναι σύντομοι. Να ξεκινήσουμε, αν συμφωνείτε, με τον κύριο Πίτε Κάρι από την Ελλάδα. Για δύο λεπτά. Κάτω από τον κύριο Μολίνα και η κυρία Καμπουθάνο και μετά οι δύο εισηγητέ του πάνελ. Κύριε Πιτικάρη, δύο λεπτά έχετε το λόγο. Ε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα λίγο παραπάνω από δύο λεπτά. Λίγο, λιγότερο, λίγο παραπάνω. Ε, οι μεγάλοι πολιτικοί ηγέτε της Ευρώπης, οι πατέρες της Ευρώπης, όταν δημιούργησαν την Ένωση, είχαν καταρχήν πίσω τους το μεγάλο βάρο ε, ε, του πολέμου, τη καταστροφή και μπροστά του το όραμα τη δημιουργία. Φτιάξαμε συνθήκε υπογράψαμε συνθήκες και προχωρήσαμε από κοινού με επιτυχία για αρκετό διάστημα. Αυτές οι συνθήκες, αυτή η νομοθεσία, το, το rule of law, ξαφνικά μέσα στην κρίση βρέθηκε να αμφισβητείται. Είδαμε ότι χώρες όπως που έζησαν την κρίση χρέους όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η, η τραπεζική κατάρρευση στην Ιρλανδία, η Ισπανία, η άδικη και πέρα από το ευρωπαϊκό δίκαιο ε, πρώτη αντιμετώπιση της Κύπρου ε, έδειξαν ότι η επίτευξη των στόχων της κοινωνικής και οικονομικής ενοποίησης δεν μπορούν να αφαιθούν μόνο στον ισχυρό συντονισμό των επιμέρους δημοσιονομικών πολιτικών. Γιατί αυτές, όπως είδαμε, είναι που να παράγουν τα χρέη και τα ελλείμματα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια νέα, μια νέα ε, οικονομική και κοινωνική και πολιτική η οποία θα βλέπει την Ευρώπη σαν σύνολο. Θα προχωρήσει στο σωστό καταμερισμό ανάλογα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε χώρα. Δεν θα τιμωρεί και δεν θα, και δεν θα δημιουργεί έτσι, δεν θα αναπαράγει μέσα από, μια ρητορική το ρατσισμό. Έχουμε μια Ευρώπη στην οποία έχουμε ρατσισμό βορρά-νότου. Απίστευτα πράγματα, αυτά θα ήταν διανόητα πριν 10, 10 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικά για την Ελλάδα και επειδή, τη ε, τη μου. Ε, η Ελλάδα όπως και ε, έζησε καταρχήν ε, την έκπτωση μιας κυβέρνησης επειδή η κυβέρνηση αυτή ζήτησε να κάνει δημοψήφισμα. Και την έζησε με πολύ έντονο τρόπο. Η Ελλάδα είδε όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα να ε, διαταράσσονται και να καταργούνται. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση τα ανθρώπινα δικαιώματα να καταστρατηγείται, όπως σας έχω γράψει στην αναφορά μου. Ε, το BBC έχει ένα άνθρωπο για τις εκλογές και γράφει ότι «If the new government η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει τις επιπτώσεις. Αυτό είπε ο Σόιμπλε. Και, ε, εκ, ε, εκβιασμών των λαών. Αυτά όμως δεν μπορούν να είναι το, το δικό μας μέλος. Ε, έχουμε στην Ελλάδα μια ταξιφόρση από τον Δόκτωρ Φως Ράχεμπαχ, η οποία δρά χωρίς να έχει κάποιο πλαίσιο εργοδοσίας χωρίς να δίνει σε κάποιο λογαριασμό, χωρίς να μας λέει με ποια διεθνή μέθοδο, με ποιο διεθνές αποδεκτό framework δρά και αξιολογεί τις δομές και ε, επιδρά στη χώρα. Το ίδιο κάνει και η Τρόικ. Ακολουθεί την πολιτική της ιστορικής υποτίμησης. Και τελειώνοντας ήθελα να σας πω ότι η καταστατήγηση των δικαιωμάτων και η πλήρης εξαθλίωση των λαών είναι του Νότου είναι ο προάγγελο τη εξαθλίωση των κρατών μελών του Βορρά, διότι στην πραγματικότητα είμαστε μια οικογένεια, είμαστε ένα οικοσύστημα οικονομιών και ανθρώπων. Η, ο φόβο, η θεωρία ότι οι λαοί του Βορρά θα αναγκαστούν να επομιστούν την οικονομική αδυναμία, δηλαδή τα δάνεια των εταίρων του, αποτελεί κατά συνθήκη ψεύδο που καλύπτει την ανυπαρξία ενό μοντέλου συνοχή και βαθέματο τη ενοποίηση αποτέλεσμα στην ανεβαρσία τη ισότιμη πρόσβαση στο κόστο χρήματο των επιχειρήσεων και του, και του τρόπου χρηματοδότηση των κρατών. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται λίγο πριν τι εκλογέ για την ανάδειξη του νέου Κοινοβουλίου, ενό Κοινοβουλίου που θα διαμορφώσει και την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από την ψήφο εμπιστοσύνη που θα χρειαστεί να δώσει στου επιτρόπου, είναι, ε, θα είναι ο ιδεολογικό προσανατολισμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ε, αν επιθυμούμε να να ξαναανακαλύψουμε μια Ευρώπη που θα ζει μέσα στη σφαίρα τη ηθική δραστηριότητα των λαών τη, που θα επαναφέρει την εθνική αξιοπρέπεια και τον εθνικό παλμό, που θα ξαναζωνέψει την ευρωπαϊκή ιδέα στι παραδοσιακέ τη αρχέ τη γεραία Υπήρου και θα διασφαλίσει την διόνυση και την αιχμή τη. Μέσα από μια τέτοια επιλογή θα ήταν δυνατόν να προσφερθεί στα κράτη-μέλη μια μόνιμη εγγύηση ελευθερία και στην Ευρώπη η στέρεη βάση για την εγγύηση του μέλλοντο του πολιτικού τη συστήματο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μπαρβαρά Μολίνα. Με δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα, σας βεβαιώνω το ότι η ανισότητα δεν είναι δευτερογενές φαινόμενο των φιλελεύθερων πολιτικών, είναι αλληλένδετες με αυτήν, είναι η ουσία των φιλελεύθερων πολιτικών. Και μια πρόγνωση. Όλα αυτά τα μέτρα λιτότητας ήδη έχουν επιπτώσεις, διότι έχουμε περισσότερες αρρώστιες, πόνο, απελπισία. Ε, βλέπουμε ότι ακόμα και η δημοκρατία υποχωρεί. Μέχρι να ανακάμψει η οικονομία, δεν θα καταφέρουν οι άνθρωποι να γίνουν καλά. Αυτοκτονούν οι άνθρωποι. Ο κύριος Αλαβράκος Ζήτησε, λοιπόν, είπα τρεις, θα τις επαναλάβω. Πρώτον, ακούστε τις κοινωνικές οργανώσεις, ακούστε τους πολίτες οι οποίοι εκφράζονται και κάνουν πολλές προτάσεις που δεν μπορώ να τις συνοψίσω βέβαια τώρα. Δεύτερον, δουλέψτε στο κοινωνικό τομέα για την υγεία. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, δηλαδή να υπάρχει δουλειά, φαΐ, στέγη, συντάξεις. Από όλα αυτά εξαρτάται η υγεία. Αν δεν υπάρχουν αυτά, κανένα φάρμακο δεν θα τα δώσει. Έπειτα, μην κάνετε τίποτα κατά της υγείας, αντίθετα, προστατεύσετε, μην μειώνετε ακόμα περισσότερο τις παροχές υγείας, αντίθετα, φροντίστε για την αγορά υγείας. Η δημόσια υγεία δεν είναι μια αγορά, είναι κάτι παραπάνω, είναι ένα δικαίωμα και είναι ένα βασικό στοιχείο του πολιτισμού που πρέπει να στηρίξουμε. Αυτό μας το διδάσκει η ιστορία. σε ευχαριστούμε κύριε Μολίνα. Μια που απευθήκατε σε μένα να σας πω ότι ναι, οι πολίτες το ξέρουν, εκφράζονται και ψηφίζουν. Όταν ψηφίζουν, ψηφίζουν κάποια, κόμματα που έχουν προγράμματα. Οπότε ο καθένας αποφασίζει τι θα ψηφίσει, στη συνέχεια οι πλειοψηφίες αποφασίζουν και οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν τα προγράμματα τα οποία εγκρίθηκαν από την πλειοψηφία των πολιτών με την ψήφο τους. Αυτό είναι η δημοκρατία. Ευτυχώς που έχουμε την τύχη και μπορούμε και ψηφίζουμε. Εντάξει, κατάλληλα για την υγεία, συμφωνώ. Τώρα, η κυρία Καπουσάνο, παρακαλώ. Όπως σας είπα ήδη νωρίτερα, θα ήταν κάτι παραπάνω από επιθυμητό και μάλιστα δημοκρατικά ανοιγκαίο, αυτοί οι οποίοι έκαναν τις απάτες σχετικά με τις προνομιούχες μετοχές να δικαστούν για την απάτη του σε βάρος πολλών πολιτών, μεταξύ άλλων και του πατέρα μου. Γιατί τότε τι παράδειγμα έχει η κοινωνία αν οι υπεύθυνοι για τις απάτες αυτές δεν τιμωρηθούν. Το έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια. Είδα ότι στη γειτονιά μου στο Ματαρό για παράδειγμα δημιουργήθηκε μια πλατφόρμα για αυτές τις προνομίφιες μετοχές και εκεί είδα τον κόσμο και τι ήταν αυτός ο κόσμος, συνταξιούχοι, ηλικιωμένοι. Δεν ήταν δηλαδή άνθρωποι που είναι επενδυτές ή που επενδύουν σε υψηλού κινδύνου επενδύσεις, όχι. Και η κατάστασή τους ήταν τραγική μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι όλη τους τη ζωή δούλευαν και τώρα τις αποταμιεύσεις τους αυτές τις χάνουν. Και μάλιστα σήμερα στην κρίση που τις χρειάζονται περισσότερο από ποτέ. Τέλος, ελπίζω του χρόνου να μην χρειαστεί να ξανάρθω για να σας πω ότι ακόμα ο πατέρας μου δεν έχει πάρει πίσω τις αποταμιεύσεις του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Καμποθάνο. Συνεπώς, ολοκληρώνεται το σημείο αυτό με τις δύο επόμενες παρεμβάσεις. Πρώτα η κυρία Θερετέλη, βέβαια και μετά ο κύριος Σερβέτο. Παρακαλώ, σας ακούμε κυρία Θερετέλη. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, δεν μπορώ βέβαια να σχολιάσω όλα όσα ακούστηκαν. Θα υπογραμμίσω όμως ορισμένα πράγματα. Κοιτάξτε, κάποιοι είπαν ότι δεν υπάρχει πολιτιστικό σοκ στην Ευρώπη. Νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση αποδεικνύει κατάφορα ότι υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση. Το κάτω-κάτω ε, καλό είναι γιατί πρέπει να γνωριζόμαστε καλό. Όσο καλύτερα γνωριζόμαστε τόσο καλύτερα θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ένα τον άλλον. Ο Γερμανός συνάδελφος αναφέρθηκε στην αλληλεγγύη και από τις δύο πλευρές. Μα έχετε δίκιο, αμοιβαία αλληλεγγύη πρέπει να υπάρχει. Συμφωνώ μαζί σας. Επιβάλλεται αλληλεγγύη. Προς κάθε κατεύθυνση ο καθένας πρέπει να βοηθάει τον διπλανό του και όλοι με κάποιο τρόπο χρειάζονται βοήθεια. Συνεπώ το είπα ότι το ευρώ όλους μας αναγκάζει να βρισκόμαστε στο ίδιο καράβι για καλό ή για κακό. Οπότε εφόσον είμαστε ενωμένοι για καλό και για κακό, δεν μπορούμε παρά να συνεχίσουμε να βοηθάμε ένα τον άλλον και να μην λέμε ότι ο βοράς έχει, είναι ο καλός, ενώ ο Νότος είναι ο κακός. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Όπως είπα και πριν σε όλα τα ζευγάρια, ακόμα και αν είναι ευτυχισμένα μεταξύ τους, πάντα υπάρχει κάποιος ε, λιγότερο περισσότερο καλό και κακό. Και η Ελλάδα, εντάξει, 2% τη ευρωζώνη είναι τη οικονομία και του χρέους. Όμω, το ελληνικό παράδειγμα διαπιστώσαμε ότι ήταν ορολογιακή βόμβα. Δεν λέω ότι οι Έλληνες έχουν την ευθύνη, πρέπει και αλλού να ψάξουμε τις ευθύνες. Και αν επιμένω γι' αυτό είναι ότι αν θέλουμε να καταλαβαίνουμε καλά ένα τον άλλον, πρέπει να αναγνωρίζουμε συγχρόνως και τι αδυναμίες μα ο καθένα. Και αυτό είναι που λέω και για την κυρία Μέρκελ, ότι φυσικά και υπάρχουν ευθύνε και πρέπει ο καθένα να αναλάβει τι ευθύνε του και ο Νότος να αναλάβει τι δικέ του βέβαια. Και οι βόρειε χώρε, πώ να το πω, είναι κάπω πιο ισορροπημένε στον κοινωνικό τομέα ή κάπω πιο λογικά διαχειρίζονται τα δικά του, αλλά οι καταστάσει διαφέρουν. Όταν πήραμε κάποιες αποφάσεις για το ευρώ, το ξέραμε. Το ξέραμε σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο Βορράς και ο Νότος. Δεν το ανακαλύψαμε προχτές. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε ότι οι Έλληνες είναι οι Έλληνες και οι Ιταλοί, α, αυτοί οι Ιταλοί είναι πάντα ίδιοι. Όχι, εντάξει μπορεί να υπάρχει διαφθορά, η μαφία κτλ. Αλλά αυτά είναι και κλισέ. Το βασικό πρόβλημα στην Ιταλία σήμερα, κατά τη γνώμη μου, ξεπερνάει κατά πολύ τα έργα σπαγκέτι western. Η, ό,τι συμβαίνει στην Ιταλία σήμερα έχει να κάνει με το σύστημα, με τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης που πρέπει να είναι αντικειμενική και να ξεπεράσει την διαφθορά. Υπάρχουν προβλήματα με τη δικαιοσύνη, με την έλλειψη ξενών επενδύσεων στην Ιταλία σήμερα. Είναι προβλήματα κατάφορα. Αλλά δεν είμαστε εμείς που θα καταλήξουμε να αποδώσουμε ευθύνε και να πούμε εμεί είμαστε οι πρώτοι στην τάξη, οι βόρειε χώρε, Όχι, υπάρχει παγκοσμιοποίηση και η παγκοσμιοποίηση απαιτεί κάποια αλληλεγγύη. Κανένας μέσα στην παγκοσμιοποίηση δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει η Κίνα ή ποιος άλλος αναδιόμενος παράγοντας. Το βασικό λοιπόν στην Ευρωζώνη και πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό είναι ότι αποτελεί μέρος της παγκόσμιας οικονομίας. Οι δικές μας οι βασικοί παράμετροι είναι καλύτεροι από αυτούς της Αμερικής ή της Ιαπωνίας. Μην αυτό Όλα θα πρέπει να τα βλέπουμε με την απόχρωση που πρέπει. Η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική όσο λέμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Θερατέλη. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Σερμπέτο. Παρακαλώ κύριε Σερμπέτο. Ευχαριστώ. Και εγώ είμαι σύντομο. Για άλλη μια φορά καταλήγουμε στα στερεότυπα και η κυρία στάθηκε στο πρόβλημα της διαφθοράς και επ' αυτού έχω να σας πω ότι όχι, εγώ δεν μπορώ να πω για τις άλλες χώρες. Μιλώ για την Ισπανία. Ζω στο Μεξικό, εκεί υπάρχει διαφορά. και στην Ισπανία σαφώς προκύπτει ότι υπάρχει μια σειρά πρακτικών παρανόμων. Εσείς λέτε ότι είναι γενική η διαφθορά. Δεν είναι κακό το ότι ανακύπτουν περιπτώσεις τέτοιες και κάποιες σύρονται συνέχεια ενώπιον των δικαστηρίων. Είναι καλό αυτό. Αυτό δεν πάει να πει όμως ότι η Ισπανία είναι διεφθαρμένη. Λειτουργεί η δικαιοσύνη. Έχουμε εκατομμύρια υπαλλήλων, λέει ο μιλής, που κάνουν τη δουλειά τους με έντιμο τρόπο. Είναι θετικό το ότι όσοι διέπραξαν απάτες πρέπει τώρα να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Βέβαια υπάρχουν προβλήματα, αυτό έφερε την απογοήτευση και τώρα τι γίνεται με την παιδεία. Πρέπει να βελτιωθεί η παιδεία στην Ισπανία. Είναι προφανές αυτό. Δεν λειτουργεί καλά. Δευτεροβάθμια παιδεία, τα πανεπιστήμια. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, αλλά πρέπει κάτι να γίνει για να λειτουργήσει όπως πρέπει η παιδεία. Και επίσης στον τομέα της ε, δημόσιας ε, υγείας. Ήμασταν περήφανοι επί δεκαετίες. Πάρα πολλοί δανείοι συνταξιούχοι ερχόντουσαν στην Ισπανία να περάσουν εκεί τον θερμό χειμώνα μας και ωφελούνται από αυτό το σύστημα δημοσίας υγείας που είναι τόσο σημαντικό να υπάρχει, αλλά θα πρέπει να σταθώ στο ότι τα πολιτικά κόμματα και οι διάφοροι φορείς δεν θα πρέπει να ευνοούν την ύπαρξη υπηρεσιών χωρίς όριο. Γιατί η κοινωνική πρόνοια κοστίζει. Και θα πρέπει τα κόμματα να πούν την αλήθεια στον κόσμο. Ότι τίποτα δεν είναι δωρεάν. Και η δημόσια υγεία επομένως απαιτεί κάποια κεφάλαια, κάποιο που να πληρώσει. Δεν θα πρέπει να κάνουν αυτήν την προεκλογική πλειοδοσία και να υπόσχονται λαού με πετραχίλια για την κοινωνική πολιτική και έτσι να μεγαλώνει το χρέος και την ύφα την πληρώνουν οι επόμενες γενιές. Κάπως καλύτερα πάντα τα πράγματα, αλλά ακόμα δεν φτάσαμε στην επιθυμητή ειλικρινία. Να ένας από τους λόγους για τους οποίους έχουμε αυτές τις επικρίσεις. Αυτό ήθελα να σας πω. Για να επιληθούν τα σημερινά προβλήματα δεν είναι απαραίτητο να φορτώνουμε τα παιδιά μας με το χρέος. Πρέπει κάποια πράγματα να διασωθούν. Και σας επαναλαμβάνω αυτό που προείπα. Η ενότητα και όχι η διάσπαση. Αυτό χρειάζεται αυτή τη ρότα πρέπει να κρατήσουμε για να βγούμε από την τρικυμία της σχέση Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο πρόεδρος. Όλους να σας ευχαριστήσω που έχετε συμμετάσχει στο πάνελ, το πρώτο πάνελ, αλλά και τους ε, αναφέροντες. Πάμε τώρα στο δεύτερο πάνελ. Πιέζει ο χρόνος. Παρακαλώ επομένω να είστε όσο γίνεται πιο σύντομοι όταν λάβετε το λόγο. Στο δεύτερο πάνελ τώρα έχουμε το βασικό θέμα, οικονομική κυβέρνηση, κοινωνική πολιτική, φορολογία, ελεγγύη, δημοσιονομικό συντονισμό. Έχουμε δύο αγορητέ. Να του καλωσορίσουμε, να του ευχαριστήσουμε που ήρθαν. Πρωτοκαθηγήτρια Ελένα Καρλέτη του Πανεπιστημίου Μποκόνια τη Φλωρεντία και την Ελένα Φλόρες. που έχει εργαστεί στην Γενική Διεύθυνση για τις Οικονομικές Υποθέσεις της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. ευχαριστώ πολύ για την ε, πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να μιλήσω για το νέο ρυθμιστικό και οικονομικό πλαίσιο. Αρχικά μου είχατε πει ότι θα μπορούσα να μιλήσω 20 λεπτά, τώρα μου λέτε 10 λεπτά. Με συγχωρείτε που θα είμαι τόσο γρήγορη. Άρα δεν θα μπορέσω να κάνω όλη μου την παρουσίαση. Βασίζομαι σε ένα βιβλίο που μόλις ε, μαζί με άλλους δύο παρουσιάζουμε ως, ε, ως ε, επιμελητές της έκδοσης. Παρακαλώ αν θέλετε περισσότερα κοιτάξτε το βιβλίο αυτό. Πολύ σύντομα να σας παρουσιάσω την οικονομική κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και μετά θα σχολιάσω δύο ε, αντιδράσεις πολιτικής, το ε, Δημοσιονομικό ε, Σύμφωνο και την Τραπεζική Ένωση. Θέλω να τονίσω τη διαφορά ανάμεσα στα μακροπρόθεσμα ε, αποτελέσματα και επιπτώσεις και τα βράχη πρόθεσμα. Είμαι οικονομολόγος, δεν είμαι πολιτικός, ούτε πολιτικός επιστήμων, αλλά θα προσπαθήσω να καταδείξω τα δημοκρατικά και κοινωνικά ε, θέματα που προκύπτουν από αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Πρώτον, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα ας δούμε το δημόσιο χρέος, τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις. Πολύ σύντομα. Αν δείτε αυτήν την εικόνα, δείχνουν τα ελλείμματα και το χρέος του δημόσιου τομέα από 1995 μέχρι 2010 και για χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία και η ε, Πορτογαλία. Δεν χρειάζεται να δείτε τις λεπτομέρειες, αλλά θα διαπιστώσετε ότι με βάση το 2008 και το έλλειμμα και το χρέος έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Πολύ πάνω από το μέσο, όρο ε, της, από το μέσο όρο της Ένωσης. Και είναι πολύ πάνω από τα κριτήρια του Maastricht το έλλειμμα είναι σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω από 20% του ΑΕΠ. Και σε ορισμένες περιπτώσεις ε, ανεβαίνει στο 120, 130, 150. Τεράστιο δημόσιο χρέος. Οι τράπεζες τώρα έχουν ε, αυξηθεί, έχουν αναπτυχθεί εκθετικά, όχι μόνο στην Ευρώπη. Αν δείτε λοιπόν ε, αριστερά σε αυτή την εικόνα, διαπιστώνετε ότι μερικές τράπεζες όπως η Deutsche Bank, η HSBC, η BNP Paribas, Credit Agricole κτλ. Και η μπλε γραμμή, η μπλε αυτή γραμμή που βλέπετε οριζόντια, δείχνουν το ποσοστό του ενεργητικού τους ως ποσοστό του ΑΕΠ, του ΑΕΠ της χώρας στην οποία βασίζονται. Βλέπετε ότι οι τράπεζες όπως η Deutsche Bank είναι 80%, 80% του γερμανικού ΑΕΠ και τράπεζες όπως η ING στην ε, Ολλανδία είναι 160% του εθνικού ΑΕΠ. Αν δείτε τώρα τις ε, ε, κόκκινες γραμμές, ε, ότι οι τράπεζες αυτές είναι πολύ μεγάλες. Δεν μπορεί λοιπόν να τις ε, σώσει ε, μια εθνική οικονομία. Ας περάσω τώρα στις επιχειρήσεις. Ποια είναι η κατάσταση τώρα. Έχουμε και δημόσιο χρέος και τέτοιες τράπεζες, τέτοιων διαστάσεων. Όλα αυτά έχουν μεγάλες επιπτώσεις στο κόστος του χρήματος για τις ε, επιχειρήσεις. Εδώ βλέπετε ε, το κόστος ε, των δανείων στην Ιταλία και Ισπανία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οι δύο κάτω γραμμές, Ιταλία, Γαλλία, Γαλλία και Γερμανία, είναι επίσης το αντίστοιχο η αντίστοιχη εξέλιξη. Από το 2010 λοιπόν υπάρχει μεγάλη απόκληση. Οι επιχειρήσει στι χώρε που έχουν πρόβλημα, όπω η Ισπανία και η Ιταλία, πληρώνουν πολύ περισσότερο από τι επιχειρήσει που βασίζονται στι ισχυρότερε οικονομικά χώρε, όπω η Γαλλία και η Γερμανία. Ξέρετε ότι υπάρχει, για παράδειγμα, ένα ε, ξενοδοχείο στο νότιο Τυρόλο που είναι στην Ιταλία και που πληρώνει πολύ περισσότερο για να δανειστεί χρήματα από ένα ε, ξενοδοχείο που είναι απλώς από την άλλη μεριά των συνόρων στην Αυστρία. Άρα είναι πολύ διαφορετικός ο ανταγωνισμός, η όρια ανταγωνισμού λόγω, λόγω του κόστους ε, χρηματοδότησης και δανεισμού. Έχουμε πρώτα απ' όλα λοιπόν το δημόσιο χρέος που σε κάποιες χώρες της Ευρωζώνης ε, είναι πολύ μεγάλο για διάφορες αιτίες. Για ιστορικούς λόγους η Ελλάδα και η Ιταλία για πιο πρόσφατους λόγους η Ιρλανδία, η Ισπανία και σε έναν βαθμό η Πορτογαλία. Υπάρχει μεγάλη διασύνδεση μεταξύ τραπεζών και δημόσιου χρέους. Ε, μολύνουν το ένα το άλλο. Και υπάρχει σοβαρή βαλκανοποίηση της ε, ενιαία αγοράς γιατί οι τράπεζες ε, δεν δανείζουν σε ξένες τράπεζες πια και οι μικρομεσαίες έχουν μεγάλο κόστος χρέωσης και υπάρχει μεγάλη μείωση της δανειοδότησης από τις τράπεζες. Άρα έχουμε αυτή την κρίση χρέους, τη χρήση ε, ε, χορήγησης πιστώσεων. Είναι λοιπόν ε, πολύ δυσχερή η κατάσταση, υπάρχει ανεργία και τρομερή ύφεση σε αυτές τις χρεωμένες χώρες γιατί έχουν υπάρξει πολλά μέτρα λιτότητας. Τώρα βέβαια οι επιπτώσεις τους είναι πολύ περισσότερο αντικείμενο συζήτηση από ό,τι στην αρχή και αυξάνεται το αίσθημα του πληθυσμού για ότι ε, ε, έχουν ε, γίνει αντικείμενο κακής αντιμετώπισης. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη οργή και απελπισία. Αλλά και στις πλούσιες χώρες αυξάνεται το αίσθημα των πολιτών δεν θέλουν να πληρώσουν για τις χρεωμένες χώρες. Τι πολιτικές υιοθετήθηκαν για να αντιδράσουν. Δύο κυρίως. Πρώτα απ' όλα το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, δηλαδή πιο αυστηρά όρια για τα ελλείμματα και το χρέος και η Τραπεζική Ένωση ο έλεγχος των τραπεζών από το εθνικό περνάει στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά υπάρχουν και άλλες μεταρρυθμίσεις που έχουν εγκριθεί ή που συζητώνται και αυτές σημαντικές. Αφορούν κυρίως τις χρηματαγορές. Η οδηγία για τις απαιτήσεις ε, ενεργητικού και ε, ρευστότητας, ούτως ώστε οι τράπεζες να είναι ισχυρότερες και επίσης περιορισμοί για τα μπόνους που πληρώνονται στις διοικήσεις των τραπεζών και για τις διαστάσεις των τραπεζών, το μέγεθος. Θα είναι αποτελεσματικές και επαρκείς αυτές οι πολιτικές. Τονίζω ότι όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις εξετάζουν τον τρόπο σχεδιασμού της Ευρωζώνης ε, πιο μακροπρόθεσμα, αλλά δεν αντιμετωπίζουν τα βράχη πρόθεσμα προβλήματα. Άρα, οι μεταρρυθμίσεις λένε, κοιτάξτε τώρα, ας επανέλθουμε σε ένα σημείο μηδέν για να αναπτυχθούμε με πιο ομοιογενή τρόπο. Αλλά υπάρχουν άμεσα προβλήματα που πρέπει να λυθούν τώρα, γιατί υπάρχει τρομερή δημόσια χρέωση, είναι πολύ ευαίσθητε τράπεζε, έχουν ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης και υπάρχει σχέση μεταξύ δημοσίου χρέου και τραπεζών. Όσο δεν αντιμετωπιστούν, δεν αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα, δεν μπορούμε να επαναφέρουμε την ενιαία αγορά, να επανέλθει η οικονομική δραστηριότητα να ε, αντιμετωπίσουμε αυτό που ο Μάριο Μόντι ε, αποκάλεσε την ψυχολογική καταστροφή της Ευρώπης. Και έτσι θα, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τα μακροπρόθεσμα προβλήματα. Λοιπόν, μακροπρόθεσμα που ακριβώς προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι πολιτικές. Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο δεν είναι και τόσο διαφορετικό από την συνθήκη Maastricht. Επιβάλλει όρια για τα δημόσια ελλείμματα και το δημόσιο χρέος. Αλλά το θεμελιώδες ερώτημα είναι θα εφαρμοστούν όλα αυτά ή όπως με το Μάστριχτ δεν θα υπάρξουν κυρώσεις για όσους υπερβαίνουν τα όρια. Το πιο σημαντικό λοιπόν είναι η Τραπεζική Ένωση, κατά τη γνώμη μου. Και γιατί, γιατί περνάει την επιτήρηση από το εθνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και γιατί όπως είδαμε οι ε, χρηματοπιστωτικές κρίσεις είναι πιο σημαντικές. Οι κρίσεις ε, στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων είναι 2-3% του ΑΕΠ, αλλά οι χρηματοπιστωτικές μπορεί να ε, ανέβουν και στο 50 και 60 και παραπάνω του ΑΕΠ, ανάλογα με το, ανάλογα με το σε πόσο επισφαλή κατάσταση βρίσκονται οι τράπεζες και επειδή είναι τόσο μεγάλες όπως είπα. Αυτά λοιπόν τα σοκ δεν μπορούν να, αντιμετωπίσουν, να τα αντιμετωπίσουν οι χώρες. Πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μπορεί η εθνική οικονομία να βοηθήσει μια τράπεζα που ε, είναι 50% του ΑΕΠ. Είναι αδύνατο. Αυτό για καθαρά οικονομικούς λόγους, ανεξάρτητα από ποιος φέρει τις ευθύνες ή άλλα θέματα κουλτούρας και νοοτροπίας. Η Τραπεζική λοιπόν Ένωση είναι μακροπρόθεσμα το πιο σημαντικό. Και πρώτα απ' όλα χρειάζεται ένας ενιαίος εποπτικός μηχανισμός που όπως είπα περνάει λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο την επιτήρηση των τραπεζών. Αυτό αποφασίστηκε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά υπάρχουν και άλλα δύο στοιχεία. Ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης, ο οποίος συζητείται έντονα, δηλαδή σημαίνει ποιος θα πληρώσει, ποιος θα βοηθήσει την τράπεζα αν έχει προβλήματα και επίσης ε, το Ταμείο για την Εγγύηση των Ευρωπαϊκών Καταθέσεων που έχει να κάνει ε, περισσότερο με τους καταθέτες. Δηλαδή ποιος θα πληρώσει τους μικροκαταθέτες αν η τράπεζα έχει προβλήματα. Αλλά αυτό ούτε καν συζητιέται αυτή τη στιγμή. Επιγραμματικά, μακροπρόθεσμα. Αν θέλουμε αποτελεσματική τραπεζική ένωση, χρειαζόμαστε και τα τρία αυτά στοιχεία. Τουλάχιστον τα δύο πρώτα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αποφασίσει να κλείσει μια Ισπανική ή Ιταλική τράπεζα και μετά το Ισπανικό κράτος ή το Ιταλικό κράτος θα πρέπει να πληρώσει για τις επιπτώσεις. Δεν έχει κάτι τέτοιο δημοκρατική νομιμοποίηση. Είναι πολύ λεπτό θέμα. Μακροπρόθεσμα λοιπόν. Ο μηχανισμός εξυγίανσης πρέπει και αυτός να περάσει στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτω ώστε να ευθυγραμμιστούν, να, να ευθυγραμμίζονται οι αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζας για ανακεφαλαιοποιήσεις με το ποιο θα πληρώσει. Και η Ευρώπη πρέπει να πληρώσει. Αλλά κάτι που με ανησυχεί πολύ περισσότερο είναι η βραχυπρόθεσμη κατάσταση. Προϋπόθεση για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και για τη χρήση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για να βοηθηθούν οι τράπεζες είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μαζί με την Ευρωπαϊκή Αρχή, Τραπεζική Αρχή να κάνουν ε, την επισκόπηση της ποιότητας του ενεργητικού και τα τεστ αντοχής για τις τράπεζες. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα εξετάσει τους ισολογισμούς των 140 τραπεζών που επιτηρεί η ΕΚΤΑΦ και ανάλογα με το αποτέλεσμα αυτής της επισκόπησης μπορεί να ζητήσει από τράπεζες να κάνουν ανακεφαλαιοποίηση. Γιατί αν δεν συμβεί αυτό, οι τράπεζες αυτές δεν θα μπορούν να ενταχθούν στον ενιαίο μηχανισμό τραπεζικής επιτήρησης. Δηλαδή, ακυρώνουμε το παρελθόν, ξεκινάμε από μια ημέρα μηδέν, όπου όλες οι τράπεζες είναι σωστά κεφαλαιοποιημένες και προχωρούμε προς το μέλλον, όπου θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους, να βοηθήσουμε τις τράπεζες που ενδεχομένως θα έχουν πρόβλημα. Λογική αυτή η διαδικασία, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Mm. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ένα δημοσιονομικό ε, ανασταλτικό μηχανισμό. Δηλαδή οποιαδήποτε τράπεζα χρειαστεί να γίνει αντικείμενο ανακεφαλαιοποίησης και θα μπορούσε να συμβεί αυτό για την Deutsche Bank. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το εθνικό κράτος θα πρέπει να παρέμβει με τον ΑΒ τρόπο και να χρηματοδοτήσει άλλη μια φορά την τράπεζα. Και πώς θα το κάνουν. Δεν μπορούν να το κάνουν. Διότι οι τράπεζες αυτές είναι πολύ μεγάλες. Δύο εναλλακτικέ λύσεις υπάρχουν. Είτε αυτή η επισκόπηση του, της ποιότητας του ενεργητικού δεν θα οδηγήσει σε τίποτα. Ή θα γίνει δηλαδή αυτό που έγινε στο παρελθόν ότι όλες οι τράπεζες περνάνε τα τεστ και αυτό βεβαίως είναι εικονική κατάσταση ή θα χρειαστούμε νέες εισρωές κεφαλαίων για τις τράπεζες και από πού θα προκύψουν. Και αυτό είναι επειδή εξετάζουμε το μέλλον με αυτό το σχεδιασμό, αλλά υπάρχει το βάρος του παρελθόντος, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Ε, ε, στην επόμενη χρονική περίοδο. Χρειαζόμαστε ένα βαθμό δημοσιονομική ενοποίηση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι στο παρελθόν ε, ήμασταν όλοι χωριστά και τώρα θα ξεκινήσουμε από κοινού. Αν εξετάσετε το βιβλίο, πολλοί οικονομολόγοι που έχουν συμβάλει με τα άρθρα του και πολλοί που διαμορφώνουν πολιτική λένε ότι χρειάζεται περισσότερη δημοσιονομική ενοποίηση πριν αρχίσει να λειτουργεί αυτό ο εποπτικό μηχανισμό για να λύσουμε τα προβλήματα τα πρόθεσμα και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο μέλλον, το μακροπρόθεσμα. Και πώς θα γίνει αυτό. Μία δυνατότητα είναι να πείσουμε τις βόρειες χώρες να χρησιμοποιήσουν τους πόρους του ε, μηχανισμού σταθερότητας ήδη, τώρα, όχι στο μέλλον, για την άμεση ανακεφαλαιοποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Είναι όμως επαρκή τα ποσά, επαρκής οι του μηχανισμού σταθερότητας. 5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, αυτές οι τράπεζες όμως είναι πολύ περισσότερο από 5% του ΑΕΠ. Μπορούμε να αρχίσουμε να, να τους δανείζουμε, να δανείζουν στα κράτη δηλαδή οι βόρειες χώρες, όχι βεβαίως ε, χωρίς τόκο. Δηλαδή θα, μπορούσαμε να, θα μπορούσαν οι βόρειες χώρες να δανείζουν ε, υποαίρεση. Δηλαδή ότι θα σας ε, χορηγήσουμε δάνεια ε, σε διάφορες δόσεις μόνο εφόσον ε, έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα μεταρρυθμίσεων και εφόσον το εφαρμόζεται. Αλλιώς επανερχόμεθα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που δίνει ρευστότητα όπως το παρελθόν. Αλλά να μην ξεχάσουμε ότι όλη η ρευστότητα που δίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ευθύνη των εθνικών κεντρικών τραπεζών. Ή υπάρχουν ε, άλλα ε, μέτρα, ε, όπως για παράδειγμα να συμμετάσχουν και οι καταθέτες στην εξυγίανση των τραπεζών. Αλλά επανερχόμεθα λοιπόν έτσι στις Ισπανικές τράπεζες που έκαναν διάφορες ύποπτες προσφορές τραπεζικών προϊόντων στους μικροεπενδυτές. Υπάρχει αυτή η σύνδεση λοιπόν μεταξύ τραπεζών και εθνικού χρέους και ε, έχει σταματήσει στην ουσία να λειτουργεί η ενιαία αγορά. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι δεν υπάρχουν ροές διαμεθοριακές. Έχουν γίνει κάποιες μεταρρυθμίσεις και μπορώ να πω ότι ε, σε σχέση με την αρχική κατάσταση έχουν γίνει ε, τρομερά βήματα προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση αλλά τώρα η εφαρμογή των μέτρων που αποφασίζονται πρέπει να γίνει με τον σωστό τρόπο και πρέπει να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις μέχρι τέλους. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει και ο μηχανισμό ε, προστασία των καταθέσεων και ο μηχανισμό εξυγεία των τραπεζών. Αλλά το πιο επίγον θέμα είναι να αντιμετωπίσουμε το βάρο του παρελθόντο για τι τράπεζε, το δημόσιο χρέο. Και αν δεν λύσουμε αυτά τα θέματα, ποτέ δεν θα λύσουμε αυτά τα άμεσα προβλήματα. Θα είμαστε κολλημένοι στα υπάρχοντα προβλήματα. Για να γίνει αυτό χρειάζεται πολύ ισχυρή πολιτική βούληση και όραμα. Και ελπίζω τώρα, μετά τι γερμανικέ εκλογέ, να ξαναξεκινήσει αυτή η προσπάθεια γιατί ήμασταν όλοι σε κατάσταση αναμονής μέχρι τις γερμανικές εκλογές. Πρέπει λοιπόν να επιτρέψουμε έτσι στην Ευρώπη και στους πολίτες να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη που είχαν στην Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο με την εμπιστοσύνη πιστεύω ότι θα ε, ε, υπερβούμε περισσότερο τα προβλήματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας, την τόσο ενδιαφέρουσα. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Λένα Φλόρες. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που μου, δίνεις, που μου δώσατε την ευκαιρία να έρθω εδώ και να συζητήσω μαζί σας κάποιες ιδέες. Και νομίζω ότι αυτά που θα σας πω εγώ είναι πάρα πολύ ωραία με την προηγούμενη παρουσίαση της κυρίας Καρλέτη. Δεν θα επαναλάβω, ε, θα προσθέσω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα από το τελευταίο σας σχόλιο, πρέπει να είμαστε σαφείς ότι οι προτάσεις που γίνονται από την Επιτροπή, από τους πολιτικούς, πρέπει να επικεντρώνονται στο τι πρέπει να γίνει τώρα. Και είναι σαφές το τι πρέπει να γίνει τώρα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε. Από πολιτικής άποψης πιστεύουμε ότι όντως θα γίνουν για την ζωτική σημασία. Πολλά λοιπόν θα θέλαμε να κάνουμε, πολλά πρέπει να κάνουμε, αλλά πρέπει να τα ιεραρχήσουμε κάπως, να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητές μας, γιατί αν δεν ξεκινήσουμε και δεν κάνουμε τα πρώτα που πρέπει να κάνουμε, τα άλλα δεν θα μπορέσουν να ακολουθήσουν, άρα πρέπει να υπάρχει συνέπεια στις προτάσεις μας. Δεύτερον, οι εξελίξεις που έχουμε για την εμβάθυνση, για την ε, ε, Δημοσιονομική Ένωση κτλ. Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα σε ένα πλαίσιο ε, χαμηλής ανάπτυξης. Είναι μια τάση που υπάρχει, δεν είναι μόνο λόγω της κρίσης. Στην Ευρώπη βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η ανάπτυξη, η δυνάμει ανάπτυξη είναι πάρα πολύ χαμηλή ακόμα και αν έχουμε ανάκαμψη, κάτι το οποίο βλέπουμε ήδη τώρα ότι ξεκινάει η ανάκαμψη. Αυτό όμως θα είναι το πλαίσιο, πράγμα που σημαίνει ότι κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα δεν είναι καινούρια, υπήρχαν ε, μπορούσαμε μέχρι τώρα μια χαρά να τα αντιμετωπίσουμε με το 2% του έπιπε κάποιος ότι είναι το χρέος, όλα αυτά θα μπορούσαν κάλλιστα να ταυτοποιηθούν. Όμως τώρα είμαστε σε, μια, σε ένα επίπεδο χαμηλό ανάκαμψης. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιο δύσκολες οι αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε και βρισκόμαστε μπροστά σε διλήμματα, αλλά έτσι είναι. Ένα τρίτο στοιχείο που θέλω να αναφέρω με ευθύ εξ αρχής και αυτό δεν είναι και με αυτό που άκουσα πριν, μερικές φορές υπάρχει σύγχυση στη συζήτηση που γίνεται ανάμεσα στο δίνω χρήματα ή δίνω δάνεια. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και μέχρι τώρα, πέρα από τα διαφορετικά ταμεία, που είναι χρήματα από τον κοινοτικό προϋπολογισμό που ανακατανέμονται υπέρ της σύγκλησης, Κατά τα άλλα, μιλάμε για δάνεια. Δάνεια που δίνονται στις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα εξυγένσης. Δάνεια είναι αυτά. Και πρέπει να είναι σαφές όταν συζητάμε με τους πολίτες και ακούμε ότι κάποιος δίνει χρήματα. Τι θα πει δίνει. Όχι. Δάνεια είναι. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Το άλλο μου σχόλιο είναι ότι σε αυτά τα πλαίσια χαμηλής ανάπτυξης, πέρα από το ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ μας, αυτό που βλέπουμε στις οικονομικές εξελίξεις και σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η διαφορά αυτή ανάμεσα στο βορρά και τον νότο δεν υπάρχει τώρα τόσο έντονη όσον αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης. Είναι και αυτή μια βασική αλλαγή. Πρέπει να δούμε γιατί. Γιατί υπήρχαν ε, κάποιες τάσεις χαμηλής παραγωγικότητας, χαμηλές εξαγωγές για τις λεγόμενες μέχρι τώρα πιο φτωχές χώρες. Ίσως είναι πράγματα που δεν ισχύουν πια. Υπάρχουν αλλαγές λοιπόν και αλλαγές βλέπουμε και σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε τις αναδυόμενες οικονομίες και τις προηγμένες οικονομίες ε, δεν υπάρχει πια αυτό το τρίγωνο των αναδυόμενων, των αναπτυγμένων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάμεσα και στις αναδυόμενες χώρες υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους. Οπότε πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο βέβαια την ΟΝΕ ναι και τον συντονισμό. Όπως είπε και, Καλέτη, και Ελένα Καλέτη, συγγνώμη, οι αλλαγές πρέπει να γίνουν. Τι άλλο. Βράχει πρόθεσμα. Έχουμε διάφορα πράγματα τα οποία αρχίζουν να λειτουργούν και είναι το αποτέλεσμα της συναπόφασης Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Έχει να κάνει με τον προπολογισμό, έχει να κάνει με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες για το μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Δεν θα λύσει την κρίση, αλλά μας αναγκάζει να δούμε και άλλα στοιχεία τα οποία είναι ζωτική σημασίας για να πετύχουμε την ανάπτυξη και την σταθερότητα στην οικονομία μας. Πολύ σημαντικό για χώρες όπως είναι η Ισπανία αλλά και άλλες που στην αρχή της κρίσης δεν είχαν δημοσιονομικό ζήτημα αλλά απέκτησαν εξαιτίας των άλλων στοιχείων στην οικονομία που ήταν αδύναμα. Συνεπώς, Έχουμε αυτά τα μέσα, εσείς συμμετείχατε εξάλλου στην διαδικασία απόφασης. Τώρα πρέπει να λειτουργήσουν όμως αυτά τα μέσα και είναι λίγο νωρί. οπότε δεν μπορούμε να πούμε ακόμα αν θα λειτουργήσουν ή όχι. Εγώ όμως ελπίζω πως ναι, γιατί είναι τόσο πολύ ανάγκη να λειτουργήσουν που θα λειτουργήσουν και νομίζω ότι όλοι οι παράγοντες, όλες τις χώρες μέλη αντιλαμβάνονται ότι αυτά τα εργαλεία τώρα πρέπει να λειτουργήσουν. Ένα άλλο στοιχείο τώρα το οποίο κάπως αλλάζει είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν με το δημοσιονομικό σύμφωνο. Θέματα συντονισμού εξάντε πολιτικής που δεν ήταν τόσο προφανή μέχρι τώρα, αλλά που μπορεί να αποτελέσουν πολύ ενδιαφέροντα μέσα για να συζητήσουμε μέτρα διαρθρωτικής πολιτικής με τις χώρες μέλη πριν καταλήξουν αποφάσεις. Και αυτό να γίνει πολυμερός, όχι μόνο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και με τις άλλες χώρες. Υπάρχει στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο λοιπόν. Εμείς στην Επιτροπή σκεφτόμαστε πώς θα γίνει αυτό στην πράξη. Μπορεί να μην χρειαζόμαστε ε, νομοθεσία. Τώρα είμαστε σε τριμερή διάλογο με τις χώρες μέλη για να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Μέχρι τα τέλη, τα τέλη της χρονιάς πιστεύω θα έχουμε μια καλύτερη άποψη για το πώς θα λάβει η χώρα ο εξάντε συντονισμός. Το θέμα είναι πάντως να συζητάμε διερθωτικές μεταρρυθμίσεις πριν αυτές αποφασιστούν. Και να μην είναι μια γενική ιδέα, αλλά να ξέρουμε συγκεκριμένα τι θέλει να κάνει κάθε χώρα και κατά πόσο αυτά συνάδουν με τις στρατηγικές και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί εδώ. Εξάντε συντονισμός λοιπόν. Φέτος για πρώτη φορά θα γίνει. Τώρα το φθινόπωρο. η άσκηση που γίνεται και με το σχέδιο προπολογισμού. Δηλαδή για πρώτη φορά, και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, για πρώτη φορά οι χώρες θα παρουσιάσουν το σχέδιο προπολογισμού τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν το υιοθετήσουν τον προπολογισμό και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γνωμοδοτήσει, θα πει δηλαδή σε τι βαθμό το σχέδιο αυτό προπολογισμού αντιστοιχεί στις συστάσεις που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη εν λόγω χώρα μέλος. Αυτή η εξάντε συζήτηση εξετάζει όλες τις χώρες, αλλά εξετάζει και τις επιπτώσεις πάνω σε ολόκληρη την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Είναι ενδιαφέρον δηλαδή να κοιτάμε τον προπολισμό της κάθε χώρας στα πλαίσια της Ευρωζώνης, δηλαδή τι επιπτώσεις θα έχει ο προπολισμός της Ισπανίας, όχι μόνο για την Ισπανία, αλλά και για ολόκληρη την Ευρωζώνη. Και τι παρατηρήσεις θα είχαμε να κάνουμε πριν υιοθετηθεί ο προπολογισμό αυτός. Η νομιμότητα λοιπόν και η λογοδοσία καταλαβαίνετε ότι είναι ζωτική σημασία. Πρέπει να πηγαίνουν εκ παραλίλου. Την ευθύνη για τον προπολογισμό την έχει το Εθνικό Κοινοβούλιο κάθε φορά, αλλά η γνωμοδότηση αυτή, η άποψη αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μετρήσει στη συζήτηση που θα γίνεται στην κάθε χώρα εν ώψη της έγκρισης του προπολογισμού της. Κοιτώντα κάπως πιο μακροπρόθεσμα τώρα. Υπάρχουν πολλά στοιχεία στο λεγόμενο blueprint, στο έγγραφο αυτό που ετοίμασε πριν από ένα χρόνο περίπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί λέμε πώς κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Και όπως ήδη υπόθηκε, Υπάρχουν ε, πολλά από τα στοιχεία αυτά ή αρχίζουν να παίρνουν σάρκα και οστά. Υπάρχουν όμως άλλα τα οποία είναι για πιο μακροπρόθεσμα. Γι' αυτά λοιπόν τα τελευταία υπάρχει ένα θέμα καθορισμού προτεραιοτήτων. Σήμερα στο πρώτο μέρος της συνεδρίασης αυτής ορισμένοι από εσά είπαν ότι υπάρχουν συστάσεις για πολιτικές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα κράτη-μέλη, αλλά ότι τα κράτη-μέλη αργούν πάρα πολύ να αποφασίσουν. Για παράδειγμα, αν έχετε ένα δημοσιονομικό στόχο και πρέπει να συμμορφωθείτε με αυτόν, ο τρόπο με τον οποίο αποφασίζουν οι χώρε να το κάνουν μπορεί να διαφέρει από τη μία χώρα στην άλλη. Αυτό το στοιχείο πιστεύω εγώ έχω ακούσει πολύ τι γίνεται στην Ισπανία, μέσα στην Ισπανία πώς τα συζητάνε αυτά τα θέματα. Αλλά πιστεύω, με πάση περιπτώσει, ότι είναι σημαντικό να συζητιέται το πώς θα γίνει αυτό, πώς θα επιτευχθεί ο δημοσιονομικός στόχος. Γιατί δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος, υπάρχουν πολλοί. Άρα λοιπόν τα κράτη πρέπει να κοιτάξουν και τα έσοδα και τις δαπάνες για να δούνε πώς θα ανταποκριθούν στο στόχο πώς θα αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές συνέπειες και πώς θα αντιμετωπίσουν την κατανομή του εισοδήματος που απορρέει από τα μέτρα αυτά. Έτσι, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Πραγματικά τα μέτρα εξυγίανσης να κατανεμηθούν δίκαια στον κόσμο. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία για το μέλλον. Εμείς στο Blueprint λέμε πώς πρέπει να έχουν οι προτεραιότητες και πώς πρέπει να εφαρμοστούν στο μέλλον, στο μελλοντικό σχεδιασμό της ΟΝΕ. Όπως είπα, η δημοσιονομική πειθαρχία έχει να κάνει με πολιτικές επιλογές. Και δύο τελευταία πράγματα που έχω να πω για την δημοσιονομική αλληλεγγύη στο Blueprint, θα δείτε ότι λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτει μια τέτοια δημοσιονομική ικανότητα. Ίσως να πρέπει να υπάρχει ένα εργαλείο σταθερότητας στην ΟΝΕ για να αντιμετωπίζονται τα σοκ και στο μέλλον. Αναφέρουμε και την ιδέα της Ελένα για τις συμφωνίες. Ίσως είναι δύσκολο να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό στην πράξη, γιατί βλέπετε αυτό που δεν θέλουμε είναι η ιδέα αυτή της ε, ε, συμφωνίας να ενισχυθεί, αλλά το σκέλος αλληλεγγύη να αποδυναμωθεί, που δεν το θέλουμε. Και σίγουρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλουμε να ανακαλύψουμε μια νέα διαδικασία. Γιατί δεν βοηθάει. Οι πολίτες δεν το θέλουν. Αν λοιπόν προχωρήσει αυτή η ιδέα, τότε οι χώρες θα πρέπει να έχουν κάποιες πολιτικές συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνες θα καθορίσουν πώς θα ανταποκριθούν, τι μεταρρυθμίσεις δηλαδή και τι πολιτικές αποφάσεις θα λάβουν. Και μετά το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, η μέρος του, θα αποτελέσει μια συμφωνία, μια σύμβαση ανάμεσα στη χώρα μέλος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά βέβαια και με χρηματοδότηση για να φανεί αλληλεγγύη. Για να υπάρχει και αυτή η αλληλεγγύη. Θα μπορούσε να λειτουργήσει και θα ήταν ένα πρώτο βήμα προς την δημοσιονομική αυτή ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα για άλλα θέματα μπορεί να μην έχουμε προχωρήσει πολύ, αλλά ίσως στους επόμενους μήνες. Πάντως, όλα εξαρτώνται από τις θέσεις των χωρών μελών. Από τις συζητήσεις που έχω ακούσει, υπάρχει φόβος, εκφράζονται φόβοι ότι θα ενισχύσουμε πιο πολύ το θέμα αυτής της σύμβασης και λιγότερο το θέμα της αλληλεγγύης. Αυτά για το που βρισκόμαστε, χωρίς να λέω ότι είναι πλήρης η παρουσίαση, αλλά θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για το ότι σεβαστήκατε το χρόνο σας. Όπως θα παρατηρήσατε έχω αναλάβει την Προεδρία. Αυτό δεν θα βλάψει το ευρώ. η κυρία Παλίνε Γκισάντα από τους νέους Ευρωπαίους Φεντεραλιστές. Παρακαλώ. Παρακαλώ ε, να είστε σύντομοι. 4-5 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε για να να σας παρουσιάσω τη θέση μας Θέλουμε να ζούμε πούμε ότι θα πρέπει να βλέπουμε την οικονομία, οι πόρους πολιτικής, οι πολιτικής επιστήμης και οι φεντεραλιστές και το διεθνές ε, κίνημα το παρουσίασε αυτό πέρσι και ζητήσαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσετε αυτές τις νέες σας αρμοδιότητες από τη Συνδίκη της Λισαβόνας για να ξεκινήσετε μια καινούργια μεταρρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να θεωρήσετε τις συνθήκες και έτσι να έχετε μια δημοσιονομική ένωση στο κοινωνικό σύστημα και κατεβάσαμε αυτή την αναφορά γιατί θεωρήσαμε ότι η διακυβερνητική συνθήκη χρειαζόταν αλλά δεν έφερε την δημοσιονομική ελληνική για να σωθεί το ευρώ και να βοηθήσει την ευρωπαϊκή Ένωση, της Ένωσης. Οπότε ε, αυτή η συνθήκη επίσης δεν έλυνε και τα προβλήματα σε σχέση με την πολιτική νομιμοποίηση. Με αυτή την αναφορά λέμε στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις αρμόδιες του, ούτως ώστε να ξεκινήσει τις, τις, ε, τις ε, για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Βέβαια, δυστυχώ δεν είναι εδώ πολλοί ευρωβουλευτέ. Ευχαριστούμε όλου όσοι ήρθαν εδώ γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί επομένω εμεί θεωρούμε ότι χρειάζεται να υπάρξει μια εκβάθρον μεταρρύθμιση. Πρώτα-πρώτα, διότι χρειάζεται ένα συντονισμό οικονομικό που έδειξε ο, μέχρι τώρα ότι αυτό χρειάζεται και έχουμε την οικονομική κρίση που, και το θέμα δεν είναι μόνο το υψηλό έλλειμμα αλλά είναι και η αντιφατικότητα το ότι έχουμε ενίο νόμισμα αλλά δεν έχουμε οικονομική διακυβέρνηση οπότε το κοινοβούλιο θα πρέπει να βοηθήσει και οι προσπάθειε που έχετε κάνει ήταν προ τα εμπρό, αλλά είδα, πάμε ότι οι συνέπειε τη κρίση πάνε πολύ παραπέρα ε, από, την, από το δευτερογενέ κοινωτικό δίκαιο και οπότε θα πρέπει να έχουμε και κάποια θεσμικά όργανα για αυτή την ε, Δημοσιονομική Ένωση. Τα είπαμε σήμερα το πρωί και εμείς ε, τονίζουμε και ανησυχούμε για το ότι η κρίση ενίσχυσε ε, τις επιφυλάξεις των Ευρωπαίων όσον αφορά την νομιμότητα την νομοποίηση της Ένωσης και όπως έχει σήμερα η θεσμική αρχιτεκτονική θα πρέπει να πάει παραπέρα από το ΑΒΕΤΟ και να έχει κάποιο ομοσπονδιακή μορφή τα είδαμε το Σεπτέμβριο του 2012, τα, τα ακούσαμε τον ε, πρόεδρο Μπαρόσο, ότι δεν έχει τα αναγκαία μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και χρειάζονται επομένω εντυπωσιακέ αλλαγέ. Στεκόμαστε επίση και στο ότι έχει περάσει η ώρα των ε, μικρών αλλαγών. Για να είναι βιώσιμη η Ένωση χρειάζεται τραπεζική ένωση, Μεσονομική ένωση και δημοκρατική διακυβέρνηση πέραν της εποπτείας χρειάζεται κάποιο ε, όργανο διεύθυνσης. Ε, επίσης ε, θα, η Δημοσιονομική Ένωση σημαίνει έλεγχο στους εθνικού προϋπολογισμούς, χρειάζεται και αρμαδιότητες ε, φορολογικές και να σπρώχνουν τα κράτη στην ανάπτυξη που έχουν πρόβλημα. Η πολιτική ένωση δεν σημαίνει μόνο να γίνεται μια σειρά συναντήσεων δημοκρατών και κυβερνήσεων, αλλά χρειάζεται πραγματικά ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και κυβέρνηση. Βεβαίω θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε από πού θα ξεκινήσουμε να βρούμε τη δημοσιονομική ελεγγύη, την Ευρωπολιτική Ένωση, αλλά είναι σαν την και το αυγό. Και τα δύο χρειάζονται για να προχωρήσουμε όπω. πρέπει. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Αυτό σημαίνει τα εξή τρία. Τραπεζική Ένωση, Δημοσιονομική και Πολιτική. Η Τραπεζική Ένωση, επαγγελματικά έχουμε πει, θα πρέπει να είναι ένα ε, πλαίσιο εγγυητικό, να χρειάζεται άμεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μέσω του Ταμείου του Ευρωπαϊκού και έτσι να συγκροτηθεί ένας φορέας εποπτείας ενιαίος στην Ευρωζώνη ε, εκεί που υπάρχουν συστημικοί κίνδυνοι και επίσης να έχουμε μια εσωτερική πλήρη αγορά στον τραπεζικό κλάδο. Η κοινή αγορά πρέπει να ολοκληρωθεί και αυτό επίσης είναι ε, η κοινή βάση για την φορολόγηση ενιαία και βελτίωση ε, όσον αφορά την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων. Επίσης, η οικονομική ε, ένωση για να είναι βιώσιμη, η Ευρώπη χρειάζεται αυτό να γίνει για να υπάρχει και κάποια πρικοδότηση, οπότε έτσι να έχουμε ε, κάποιους φόρους που να προέρχονται τα κράτη-μέλη και έτσι να αυξηθεί η αξιοπιστία του ενιαίου κοινού νομίσματος να έχουμε και τα project bonds και τα, και τα ευρωομόλογα, ούτω ώστε να μπορούμε να έχουμε επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να ελκύσουμε επίσης επενδύσεις ε, απ' έξω αλλά και από το της Ένωσης και έτσι να υλοποιήσουμε τη στρατηγία το 2020. Γι' αυτό και είπαμε έχουμε το 2020 για να έχουμε σε ενέργεια, μεταφορές και τηλεπικοινωνίες επενδύσεις πρέπει όμω κάτι να κάνουμε επίση για να έχουμε περισσότερη δημοσιονομική ελεγγύη. Οπότε χρειάζεται να κινηθούμε προ κάποιο είδου ε, κατανομή του κρατικού χρέου. Ε, και σε αυτό βοηθούν τα ευρωομόλογα, αναδιανομή του κόστου του δανεισμού και να βοηθήσουμε τα πιο αδύναμα μέλη της Ευρωζώνης, να το τα βοηθήσουμε να έχουν πάλι ανάπτυξη και αντιμετωπιστεί η το, το credit crunch τέλο πάντων η, το πρόβλημα της ρευστότητα. Οπότε έτσι θα αυξηθεί η νομοποίηση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μόνο η διακυβερνητική συνεννόηση δεν μπορεί να αποκαταστήσει ε, αυτήν την ένωση και χρειάζεται επομένως η Πολιτική Ένωση για να έχουν την νομιμοποίηση τα θεσμικά όργανα και ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός να έρθει στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακόμα χειρότερα, έχουμε τις πρόσφατες αποφάσεις που έχουν περιθωριοποιήσει τα πραγματικά υπερεθνικά οργανώματα στο το Κοινοβουλίο. Μόνο έτσι μπορεί να έχουμε μια συνεκτική πολιτική. Να υπάρχει ένα Υπουργείο Οικονομικών Ευρωπαϊκό να λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο και να εκπροσωπεί στο Δουνουτού, στην Παγκόσμια Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, μόνο μια κοινή δημοσιονομική πολιτική, οικονομική πολιτική κοινή στις χώρες της Ευρωζώνης πρόκειται να βοηθήσουν τόσο ώστε να σταυροποιηθούν οι αγορές και να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων. Δεν ξέρω τώρα είναι η κατάλληλη ώρα, γιατί ορισμένοι λένε ότι θα έχουμε μια πολιτική κρίση που θα έρθει να προσθεθεί στην οικονομική κρίση αν έχουμε τέτοιε μεταρρυθμίσει. Δεν μπορούμε ποτέ να ξέρουμε ποιο είναι το τέλειο χρονικό σημείο. Όμω το 2014 έχουμε το μεγάλο οικονομικό ραντεβού για τι ευρωεκλογέ. Οπότε δίνεται η ευκαιρία να λάβουν τι ευθύνε του τα πολιτικά κόμματα και όλοι οι υποψήφοι, ούτω ώστε να μπορέσουν να εξηγήσουν το όραμά του για, για την εντολή που θα αναλάβουν και έτσι να υπάρχει αλληλεγγύη των λαών και να βοηθήσουν, όπως λέει το πρωί της συνθήκης, στην οικονομική πρόοδο και έτσι να βρεθεί το αδιέξοδο από την κρίση. Ήρθε η ώρα, υποψήφιες ευρωεκλογέ, αλλά και τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να προσφέρουν τις προτάσεις τους για τη μεταρρύθμιση του πολιτικού συστήματος. Του χρόνου αυτό θα είναι μια ευκαιρία με τις ευρωεκλογέ να γίνει μια τέτοια συζήτηση με ευρωπαϊκή διάσταση, μια που πιέζει ο χρόνος τονίζουμε ότι είναι μεγάλη αυτή η πρόκληση. Πρέπει επομένω να δούμε τι αλλαγέ χρειάζονται και αυτό θα πρέπει να γίνει με διαβούλευση, με προβληματισμό, με συμμετοχή των Ευρωπαίων. Γι' αυτό και για μα χρειάζεται να υπάρχει μια συντακτική συνέλευση μετά τι εκλογέ, με, μετά τα όσα για τι εκλογέ και έτσι οι επόμενες φάσεις της ολοκλήρωσης θα πρέπει να γίνουν με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων, με τους προσώπους τους, τα κοινοβούλια τα εθνικά, το ευρωπαϊκό και τις κοινωνίες των πολιτών. Και έτσι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε, να βελτιώσουμε τις συνθήκες, όχι με συναντήσεις κορυφής, αλλά μια τέτοια συλλεκτική συνέλευση. Ευχαριστώ. Πολλές προτάσεις για το κοινοβούλιο μας, για τους συναδέλφους. Ίσως λοιπόν ορισμένες ε, ομάδες να μπορέσουν να αναλάβουν αυτές τις ε, προτάσεις να τις κάνουν δικές τους. Πρώτα απ' όλα λοιπόν έχουμε μία αναφορά για προσβολή μέσω της Τρόικα ε, και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Κομισιόν του κυρίου Πιτικάριου, που έχει το λόγο. Τρία λεπτά παρακαλώ. Ε, οι μεγάλοι πολιτικοί ηγέτες της, ε, η Ευρώπη είχε την ευκαιρία να έχει πολύ μεγάλου πολιτικούς ηγέτες τον Ζισκάρντε Στέν, τον Χέλμουντ Σμιθ, τον Ζακ Τελόρ, τον Κωνσταντινό Καραμαλή από την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι από τα μέλη, από τα πρώτα 12 μέλη της ΕΟΚ, ε, τον Χέλμουντ Κόλ, ανθρώπους με τεράστιο πολιτικό βάρος που κατάφεραν και προώθησαν την Ευρώπη προς μια ενότητα. Όμως Παρά το δικό του πολιτικό βάρο, είδαμε ότι οι συγκρούσει των εθνικών συμφερόντων απαιτούν να υπάρχει επιμονή και υπομονή προς τον δρόμο για μια ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Έγινε από νωρίς κατανοητό ότι η πολιτική ενοποίηση είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής δυναμικής, των κοινωνιών που θα είναι έτοιμες να ενοποιηθούν. Έτσι προτάθηκε να προηγηθεί η οικονομική ενοποίηση με κύριο όχημα ένα κοινό νόμισμα. Έγινε πιστευτό ότι τα ωφέλη από την ανάπτυξη, τη σταθερότητα του νομίσματο, η ελευθερία κίνηση κεφαλαίων και ανθρώπων και η σταδιακή προσαρμογή του προ τα πανευρωπαϊκά ιδεώδη θα προέκυπταν σχεδόν αυτόματα και τελικά θα κατορθώναμε να ενοποιήσουμε πολιτικά, δηλαδή να δημιουργήσουμε μια συνομοσπονδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί είπαν μάλιστα ότι ένα τέτοιο περίπου πείραμα έγινε και στην Ανατολική και η Γερμανία κατά την Ένωση. Και θα μπορούσε ίσω να είναι και ο δρόμο για την δική μας πορεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από νωρί είχε ανακαλύψει ότι υπάρχουν, είχε, είχε διαγνώσει την ανάγκη ανακύκλωση των πλεονασμάτων. του. Είχαμε τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, όπου λεγόταν πακέτα Ντελορένα, 2, ε, το τρίτο κοινωνικό πλαίσιο στήριξη, το, το, νέο, το νέο πλαίσιο στήριξη. Η πολιτική απόφαση των κυριαρχών κρατών να περιορίσουν τι εξωστατικέ πολιτικέ οδήγησε το δικοδόμημα του ευρώ σε ένα κρίσιμο σημείο. Η πορεία των πραγμάτων απέριξε πω χωρί την ύπαρξη συνεπού συνευτικού προγράμματο οικονομική σύγκληση, ενό προγράμματο οργανική ενότητα τη ευρωπαϊκή οικονομία, στηριζόμενο σε συμπληρωματικέ οικονομικέ πολιτικέ και ευρωπαϊκό καταμερισμό, η οικονομική ενοποίηση είναι ένα ανέφικτο στόχο. Το βλέπουμε αυτό σήμερα μέσα από τη διεύθυνση των πλεονασμάτων και των ελλημάτων, των εμπορικών πλεονασμάτων και των εμπορικών πλεονασμάτων. Η κρίση χρέου στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, την Ισπανία, η τραπεζική κατάρρευση τη Ιρλανδία και τα προβλήματα που προέκυψαν στην Κύπρο απέδειξαν ότι η επίτευξη των στόχων τη οικονομική γενική νομοποίηση δεν μπορούν να αφαιθούν μόνο στον ισχυρό συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών, όπω ισχυρίζεται η Επιτροπή. Ε, το, το, ΠΑΚ είναι μία πρόταση η οποία είναι στα όρια τη νομιμότητα μια και η Επιτροπή αποκτά αρμοδιότητες που, δεν προέρχονται από το υπέριο των λαών. Γιατί το υπέριο, την εξουσία την έχουν οι λαοί και δεν το έχουν αυτή τη στιγμή με κάποιο τρόπο μεταφέρει στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεν εκλέγεται και όλα. Η Νομισματική Ένωση είναι μια με οποία, εφόσον δεν εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση και το επαρκέ επίπεδο στο κόστο χρήματο των επιχειρήσεων. Βλέπουμε επιχειρήσει από τον Νότο να αναγκάζονται να μεταφέρουν την έδρα του στι χώρε του Βορρά. Πρόσφατα στην Ελλάδα είχαμε την ε, η Βιοχάλκο, η οποία πήγε στο, ήρθε στο βασίλειο του Βελγίου προκειμένου να μπορεί να, να βρει χρηματοδότηση. Δεν υπάρχουν πόλει, δεν μπορούν οι επιχειρήσει στον Νότο να, βρουν, να έχουν πρόσβαση στην τραπεζική αγορά, στη ρευστότητα. Είναι σημαντικό να θεσμοθετήσουμε την κυριαρχία των ανθρώπινων αξιών επί των οικονομικών συμφερόντων. Άλλωστε, είναι αδιανόητο να θεωρούμε τη φοροδιαφυγή, όπω είπε και η κυρία Ευρωβουλευτή, ω επέσχυντο κοινωνικό και οικονομικό έγκλημα, αλλά την ίδια στιγμή, λόγω έλλειψη μηχανισμού ελέγχων αλλά τη συνεκτικότητα που έχουμε επιδείξει να επιβραβεύουμε τη φοροαποφυγή διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών μέσα από τα διάφορα μικρά ή μεγάλα παραθυράκια. Όπω είναι η offshore. Τέλο, δεν είναι κατανοητό για ποιο λόγο δεν υπάρχει δημοκρατικό έλεγχο και λογοδοσία τη Κεντρική Τράπεζα. Η Κεντρική Τράπεζα σε ποιο Δεν λογοδοτεί, δεν στο Κοινοβούλιο δεν λογοδοτεί ε, και υπάρχουν μάλιστα και κεντρικές τράπεζες χωρών κρατών μελών που την πλειοψηφία των μετοχών τον έχουν, την έχουν οι ιδιώτες, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα. Και μάλιστα αυτό συμβαίνει την ώρα που θέλουμε να θέσουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως πυλώνα, ως, ως watchdog της ε, ε Τραπεζικής Ένωσης. Η μη επίτευξη του στόχου τη ευρωπαϊκή οικονομική και κοινωνική ενοποίηση δεν αποτελεί ατύχημα, αλλά συνέπεια τη κυρίαρχη οικονομική πολιτική που ακολουθήσαμε ω σήμερα. Η ίδρυση μηχανισμού χρηματοπιστωτική σταθερότητα, το οποίο τα μέλη από την ιδρυτική συνθήκη απολαμβάνουν ασυλία έναντι κάθε άλλη αρχή, προσβάλλει την αρχή τη λογοδοσία του accountability. Δεν ναι. είναι δυνατόν να λέμε ότι θα έχουμε δημοκρατία και θεσμού όταν Υπάρχουν οργανισμοί των οποίων τα μέλη δεν έχουν λογοδοσία. Κύριε ε, θα πρέπει παρακαλώ να πείτε μόνο μία φράση. Μία φράση παρακαλώ. Για τον επόμενο μετά. Δεν είναι το, το Άγιο Σκοποτήρου. Άλλωστε στην η Ελλάδα δανείστηκε περίπου 200 δισεκατομμύρια για να σώσει 160 δισεκατομμύρια καταθέσει. Ε, είναι που είναι το Άγιο Δισκοπότητο είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο νόμος, η πολιτεία, ο πολιτισμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Äh, Ωραία, πολύ καλή φράση για το τέλος. Η επόμενη αναφορά του κυρίου Βούκ για την χρηματοπιστωτική κρίση. Ο κύριος Βούκ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Πριν έρθω, μου είπαν να ετοιμάσω την ομιλία μου, να σας τη δώσω, το έκανα. Αλλά θέλω να σχολιάσω και μερικά πράγματα που ακούστηκαν εδώ σήμερα, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό. Ακούσαμε για τον αγώνα μεταξύ Βορρά και Νότου. Εγώ έρχομαι από τον Νότο, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι δεν συμφωνώ με αυτά που άκουσα πριν για την αντιπαράθεση αυτή ανάμεσα στο Βορρά και στο Νότο. Στο Νότο το ποσοστό οργανωμένου εγκλήματος των λευκών κολάρων είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στο Βορρά. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Νότια Ευρώπη. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς το πρόβλημα, η διαφθορά δηλαδή και το οργανωμένο έγκλημα είναι που τελικά καταστρέφει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, πρέπει πολύ προσεκτικά να ψάξουμε για τη λύση. Είμαι από τη Σλοβενία και τέτοιου είδους εγκλήματα είναι αρκετά διαδεδομένα. Ορισμένοι λένε ότι πρέπει να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί φοβούνται ότι κάποια μέρα θα υπάρξει κράτος δικαίου στη Σλοβενία και όλα αυτά που κλέβανε θα τα χάσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσει μια πολιτική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκρήματος, μια ευρωπαϊκή FBI, δεν ξέρω. Γιατί όταν βλέπω την κατάσταση στην Σλοβενία δεν έχει λύση. Κανείς μέσα από τη Σλοβενία δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα γιατί όλα είναι στα χέρια αυτονών. Η γεωπολιτική, η πολιτική, η δημόσια δίκηση, τα μέσα ενημέρωσης, η δικαιοσύνη, τα πάντα είναι στα χέρια αυτονών των λευκών κολάρων. Και προφανώς το ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία κτλ. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ πιστεύω ότι πρέπει πολύ σοβαρά να εξετάσει αυτό το πρόβλημα. Αν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάψει να εφίσταται κάποια στιγμή. Και τώρα έρχομαι στην αναφορά τη δικιά μου. Από ό,τι φαίνεται, ο πολιτισμός μας, τουλάχιστον του δυτικού κόσμου, έχει αποτύχει να λύσει το πρόβλημα της ρευστότητα. Τα χρήματα είναι ένα δημόσιο αγαθό που επιτρέπει την, ε, τις συναλλαγές, την ανταλλαγή προϊόντων και λειτουργία της οικονομία. Όμως, ανάλογα με το τι χρήμα κυκλοφορεί, εξαρτάται ο τρόπος ε, με τον οποίο γίνονται οι ανταλλαγές αυτές, πώς συλλέγονται οι φόροι κτλ. Αν τα χρήματα που κυκλοφορούν δεν αρκούν, τότε μειώνεται το ΕΠ, αυξάνεται η ανεργία και τα έσοδα από τους φόρους μειώνονται, ενώ οι δημόσιες δαπάνες αυξάνουν. Είναι προφανές λοιπόν ότι η δημοσιονομική πολιτική, η οικονομική πολιτική είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της εθνικής οικονομικής πολιτικής. Ποιος όμως την καθορίζει αυτή την νομισματική πολιτική? Καθορίζεται από το αυτόνομο δημοσιονομικό σύστημα. Οπότε το ερώτημα είναι, τα συμφέροντα δημοσιονομικού αυτού συστήματος συνάδουν με τα συμφέροντα του κόσμου. Η απάντηση είναι όχι και πάλι όχι. Αυτό ακριβώς δείχνει ποια είναι η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωζώνη εδώ και χρόνια βρίσκεται σε κρίση. Η οικονομική ανάπτυξη είναι πολύ χαμηλή, η ανύπαρκτη, η ανεργία είναι υψηλή και αυξάνει, το δημόσιο χρέος αυξάνει, επειδή αυξάνουν και οι κοινωνικές δαπάνες και το χρέος του ιδιωτικού τομέα επίσης αυξάνει. Όλη η δημοσιονομική και οικονομική κατάσταση τελικά είναι σχεδιασμένη για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του τραπεζικού λόμπι. Το ίδιο ισχύει και στι ΗΠΑ, όπου έχουν 17-3 δολάρια ε, χρέο, το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να πληρώσουν. Είναι προφανές ότι κάτι δεν πάει καλά με τη ε, δημιουργία χρήματο μέσω του χρέους. Όταν το οικονομικό σύστημα και οι τράπεζες χρησιμοποιούν τελικά παραστατικό χρήμα από το τίποτα. Η πιο σημαντική αιτία της οικονομικής κρίσης είναι ότι τα χρήματα μπαίνουν στη κυκλοφορία ως ε, χρέος και τελικά ο δημόσιος τομέας, ο ιδιωτικός τομέας και τα νοικοκυριά δεν επωφελούνται το, το χρέος αυτό κληρονομιέται στους επόμενους και δεν αποπληρώνεται ποτέ. Αυτή είναι και η ουσία του τραπεζικού συστήματος. Οπότε το ζωτικό ζήτημα εδώ είναι ποιος είναι τελικά ο πιστωτής και ποιος είναι αυτός που πληρώνει. Τελικά ο δημόσιος τομέας είναι αυτός ο οποίος χρεώνεται, ενώ οι τράπεζες είναι αυτές που παίρνουν τα χρήματα. Ενώ θα έπρεπε να ήταν το αντίθετο, η νομισματική πολιτική θα έπρεπε να γίνεται έτσι, όπου να αποφελεί το δημόσιο τομέας. Πώς να το αλλάξουμε αυτό όμως όταν οι τράπεζες αυτές που δημιουργούν και την οικονομική κρίση και την νομισματική κρίση και την ανεργία κτλ. Όλα αυτά δεν είναι προς το συμφέρον του κόσμου, των κυβερνήσεων, ε, των λαών, όχι είναι υπέρ του τραπεζικού συστήματος. Και γιατί, διότι οι εμπορικές τράπεζες κατά τη διάρκεια της κρίσης καταφέρνουν να αγοράζουν φτηνά γη, ακίνητα ή και τίτλους και επιπλέον κερδίζουν φοβερά χρήματα δανείζοντας το δημόσιο τομέα ο οποίος αντιμετωπίζει δυσκολίες και μειώνουν τη ρευστότητα η κρίση τελικά είναι χρυσορυχείο για τις τράπεζες. Οι πλούσιοι τραπεζίτες έχουν γίνει πιο πλούσιοι και οι φτωχοί έχουν γίνει πιο φτωχοί. Πώς να αλλάξουν όλα αυτά. Η πολιτική του δημοσικού συστήματος πρέπει να βγει από τα χέρια του λόμπι των τραπεζών και πρέπει να πάει στα χέρια των αρχών, των εθνών και των κυβερνήσεων. Το ωφέλη από την έκδοση παραστατικού χρήματος πρέπει εν μέρει τουλάχιστον να πηγαίνει στο δημόσιο τομέα και όχι μόνο στο τραπεζικό λόντι οι χώρες θα πρέπει να μπορούν να έχουν ένα δίκαιο μερίδιο ε, στο χρήμα αυτό ετησίως, κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να τους χρεώνεται ως χρέος. Έτσι θα μπορούν να αποφύγουν την υπερβολική χρέωση των χωρών και του δημόσιου τομέα. Το αρχικό δικαίωμα για παραστατικό χρήμα είναι δικαίωμα του κράτους και όχι ενός αυτόνομου δημοσιονομικού συστήματος, το οποίο τελικά γίνεται ένα οικονομικό παράσιτο το οποίο υποφελείται όλο και περισσότερο από μερίδιο του ΑΕΠ. ΑΕΠ το οποίο κανονικά ανήκει στις χώρες και στους λαούς. Και γι' αυτό είναι εσφαλμένη η πολιτική λιτότητα. Σε ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ για τις εξηγήσεις σας αυτές. Τώρα. Μέχρι τις 12.45 θα έχουμε τους διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος, και υπάρχουν τρεις ακόμα συνάδελφοι οι οποίοι θέλουν το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ να περιοριστείτε 35 λεπτά το πολύ ο καθένας. Για να μπορέσουμε και να συζητήσουμε μετά. Παρακαλώ. Ο κύριος Λάινεν πρώτα. Να αρχίσετε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα, θα σας δώσω ένα κείμενο με τα όσα έχω να δηλώσω, αλλά έχω να πω επιγραμματικά τα εξή ότι θα πρέπει να δούμε το ότι τα δικαιώματα των πολιτών καταπατούνται όσον αφορά την οικονομική κατάσταση και με χαρά μου βλέπω ότι η Επιτροπή των Αναφορών το θέμα αυτό το έχει πάρει πολύ στα σοβαρά και έχουμε τώρα τους ε, προσώπους των πολιτών, εμάς, δηλαδή που θα πρέπει να υπεραμεινθούν των πολιτών. Και επομένως δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω ε, με όλα όσα είπε η Πολύν Ζεσόν για το ότι έχουν πληγεί κυρίως οι νέοι από αυτή την ε, κρίση. Για να βγούμε από την κρίση πρέπει να δώσουμε μια προοπτική στους ανθρώπους. Το κοινοβούλιο μας λοιπόν πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία ούτως ώστε να ε, διαμορφωθεί αυτή η προοπτική. Όπως ε, ξέρετε, στη Γερμανία μόλις έληξε η προεκλογική εκστρατεία, την επόμενη Κυριακή έχουμε εκλογές στην ε, Αυστρία. Από καθαρά εθνική προοπτική συζητούν όλοι για την Ευρώπη. Δεν έχουμε λοιπόν ένα ευρωπαϊκό επίπεδο για την κοινή συζήτηση για όλους μας. Για τα προβλήματα αλλά και για τις λύσεις τους. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η πρόταση να κάνουμε μια τρίτη συντακτική συνέλευση ε, αμέσως μετά τις επόμενες ευρωεκλογές, ούτως ώστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο όλα τα κοινοβούλια, οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχεδιάσουν την επόμενη φάση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και να την προετοιμάσουν. Αυτή η συντακτική συνέλευση πρέπει να είναι ανοιχτή, διαφανής, με συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, με τα σχόλια και τις προτάσεις τους. Σύντομος λοιπόν, χρειαζόμαστε περισσότερη, όχι λιγότερη Ευρώπη. Ε, η ΟΝΕ ναι, έχει μόνο ένα πόδι, χρειάζεται ένα δεύτερο πόδι, η Οικονομική και Χρηματοπιστωτική Ένωση σε τελευταία ανάλυση θα πρέπει να γίνει όπως και αν την αποκαλέσουμε πολιτική ένωση. Χρειαζόμαστε περισσότερους μηχανισμούς αλληλεγγύης, χρειαζόμαστε περισσότερη δημοκρατία. Χρειαζόμαστε δημοκρατικό έλεγχο της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής και όχι μόνο εκτελεστικό φεντεραλισμό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή ακόμη χειρότερα μέσω μιας ε, τρόικα που κανείς δεν ε, έχει εκλέξει και κανείς δεν μπορεί να, ε, κανείς δεν μπορεί να ελέγξει και να, είναι υπόλογη. Πρέπει λοιπόν να είμαστε απόλυτα σαφείς, να στείλουμε σαφές μήνυμα και στους συναδέλφους μας στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και στους πολίτες ότι θέλουμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά τους και επιδιώκουμε να βρούμε τρόπους για να εγγυηθούμε και στο μέλλον τα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Γιολάινεν. Ο Άντζο Νταφ, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα το πρωί. μάθαμε για τα απτά αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης σε διάφορα κράτη-μέλη. Και ο τρόπος διαχείρισης ε, της κρίσης ε, που ε, εφαρμόσαμε τα τελευταία πέντε χρόνια, συμφωνώ ότι αύξησε τον τεχνικό, τεχνοκρατικό χαρακτήρα της ενωσιακής διακυβέρνησης. Υπάρχουν πολλοί πολιτικοί που εξάγουν το πόρισμα από αυτήν την διαχείριση της κρίσης ότι πρέπει να επαναπατριστούν αρμοδιότητες από την Ένωση προς τα κράτη-μέλη και να ενισχυθεί η εξουσία των εθνικών κυβερνήσεων, κοινοβουλίων, τραπεζών, δικαστηρίων επί της οικονομικοπιστωτικής διαχείρισης της ενωσιακής πολιτικής. Διαφωνώ κάθετα με μια τέτοια προσέγγιση. Το αντίθετο πιστεύω ότι χρειαζόμαστε. Ό,τι δηλαδή Η εκτελεστική μας εξουσία έχει αρκετά κατακερματισμένες αρμοδιότητες. Διάσπαρτες ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διάφορους εποπτικούς μηχανισμούς κτλ. Όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της δημιουργίας μιας ισχυρής ομοσπονδιακής διακυβέρνησης της Δημοσιονομικής Ένωσης. Και μου προκαλεί αισιοδοξία η συζήτηση που κάναμε εδώ. Επίσης, μου προκαλεί ενδιαφέρον αλλά και απορίες ε, η πρόταση του Προέδρου Μπαρόζο να δημοσιεύσει βασικές αρχές για την Οικονομική και Πολιτική Ένωση πριν τη λήξη της θητείας του Κοινοβουλίου. Ελπίζω η Επιτροπή και τα πολιτικά κόμματα με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουν να υπάρξει μια πιο σοβαρή και στόχο προσιλωμένη πολιτική συζήτηση κατά την προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογέ. Πολύ λοιπόν πιο έντονη από ό,τι είχαμε μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τελευταίος, ο Στάθμος Χέφνα. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε πολλά σήμερα για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Γιατί οι πολίτες μας ε, έχουν ε, θυγεί ιδιαίτερα. Και συζητάμε και πώς λοιπόν θα εφαρμόσουμε ο μεγάλος Γκέτε είχε πει ότι πιο σημαντικό από το τι είναι το πώς θα το εφαρμόσουμε. Γι' αυτό χαίρομαι που στο κέντρο των συζητήσεών μας έχουμε αυτό το θέμα. Γιατί υπάρχουν δύο οδοί. Από τη μία να παρατηρήσουμε αμέτωχοι ότι υπάρχει όλο και περισσότερη επαναθνικοποίηση της ε, λήψης αποφάσεων. Είναι καθαρά τεχνοκρατική η αντιμετώπιση της πολιτικής από, κάτω, συγγνώμη, από πάνω προς τα κάτω και οι πολίτες είναι απλώς παρατηρητές, δεν παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικής. Και γι' αυτό θεωρώ ότι εδώ είναι το κλειδί θα μπορέσουμε να υπερβούμε την κρίση, διότι η κρίση δεν είναι μόνο τεχνικού τύπου κρίση, είναι πολύ βαθύτερα κρίση, επειδή οι πολίτες διαρωτώνται δικαιολογημένα για ορισμένα θέματα και δεν λαμβάνουν απαντήσεις. Προς ποια κατεύθυνση θα προχωρήσει η Ευρώπη, τι εννοούμε ατομικές ελευθερίες, πώς τις συνδυάζουμε με την αλληλεγγύη και την κοινωνική ευθύνη ε, στο οικονομικό μας πλαίσιο. Πώς θα τα φέρουμε αυτά σε πέρα στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε από τη μία σταθερότητα, αλλά από την άλλη αλληλεγγύη. Πρέπει να το συζητήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσο εμένουμε σε εθνικές συζητήσεις, δεν θα υπάρξει περισσότερη ενοποίηση. Αντίθετα, περισσότερος κατακαιρματισμός. Γιατί η επανα, επανεθνικοποίηση σημαίνουν ε, η επενθυνικοποίηση. λοιπόν αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες κάθε χώρα λένε όχι μας ενδιαφέρει μόνο τι θα κάνουμε εμεί για τη χώρα μας, τι θα κάνει η κυβέρνησή μας. Μόνο από κοινού θα υπερβούμε την κρίση. Για την Ευρώπη αυτό σαφώς σημαίνει ότι πρέπει να αποκτήσουμε και άλλα εργαλεία. Ήδη τα ανέφεραν ορισμένοι, δεν θα επαναλάβω, αλλά θα το επιτύχουμε μόνο εάν οι συνθήκες μας που περιέχουν πολλά σημεία που είναι πολιτικά αναγκαία, αλλά δεν τα περιέχουν όλα. Πρέπει όμως να περιλάβουν και πολύ πιο συγκεκριμένα μέσα, εργαλεία, άρα πρέπει να εξελιχθούν περαιτέρω. Η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει διαδικασία για αυτήν την αναθεώρηση. Δηλαδή να υπάρξει μια Ευρωπαϊκή Συντακτική Συνέλευση. Εγώ νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πραγματικό σημείο καμπής για την Ευρώπη. Διότι για μεγάλο χρονικό διάστημα η μεταρρύθμιση των συνθήκων ήταν μόνο θέμα κυβερνήσεων. Εάν γίνει μεταρρύθμιση μέσω συντακτική συνέλευση θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση στην Ευρώπη με του πολίτε. Δεν έχω χρόνο για να πω πολλά. Γιατί για μένα το θέμα είναι πώς θα συμμετάσχει η κοινωνία των πολιτών. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Πρώτον, η συνέλευση αυτή, όπως προβλέπουν οι συνθήκες, Πρέπει να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει δημοκρατικά. Δεν αποκλείουν οι συνθήκε, ένα τμήμα των συμμετεχόντων να εκλεγούν απευθεία από τους πολίτες. Δεύτερον, η κοινωνία των πολιτών μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία. Δηλαδή, ας πούμε, αν έχουμε 100.000 πολίτες που να κάνουν μια συγκεκριμένη πρόταση, τότε να την αναλάβει και να τη συζητήσει αυτή την πρόταση ε, η συνέλευση. Τρίτον, χρειάζεται χρόνο η συνέλευση για να συζητήσει αναλυτικά και να μην υποβάλει τις προτάσεις της σε μία, σε μία, στις κυβερνήσεις μόνο, αλλά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, για να μπορέσουν όλοι να συζητήσουν, να μπορέσουν περαιτέρω να επεξεργαστούν και μετά να το υποβάλουν στους πολίτες της Ευρώπης προς έγκριση. Θα ήταν πραγματικό σημείο καμπής, ουσιώδης αλλαγή. Έτσι θα καταλάβουν ότι η Ευρώπη δεν είναι κάτι μακριά από αυτούς, η Ευρώπη είμαστε εμείς εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το πεπρωμένο της Ευρώπης και με αυτήν την νέα δημοκρατική αλληλεγγύη θα συμμετάσχουμε όχι μόνο ως κυβερνήσεις αλλά οι ίδιοι πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Χέφνερ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Διότι δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος. Δύο λεπτά. Να μας πείτε τι θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Στραβελή και ονομάζομαι και ασχολούμαι με την πληροφορική. Και έχω δύο πάρα πολύ σύντομε ερωτήσει. Η προφορική σχέση με την ιατρική. Πώ μπορούμε να τροπήσουμε μια ευρωπαϊκή συνθήκη μέσω ε, ε, πρωτοβουλίων των Ευρωπαίων πολιτών. Δηλαδή είναι θέμα μεθοδολογικό. Πώ μπορούμε να αντικαταστήσουμε την Τρόικα με κάποια άλλη μέθοδο και να βοηθήσουμε τι χώρε εκείνες που έχουν πληγεί πολύ από την κρίση. Φερρυπίν. Πρώτον κάτι σαν το σχέδιο Μάρσαλ εκείνο το οποίο επικαλέστηκαν οι Αμερικανοί μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και απέδωσε αποτελέσματα πολύ καλά. Τελευταία με ερώτηση. Οι ειδικοί είναι πάρα πολύ απεσιόδοξοι. Μιλάνε για πάνω από 20 εκατομμύρια Ευρωπαίων οι οποίοι πρόκειται να φτωχύνουν ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Και σε ρωτώ, τι λογαριάζεται να κάνετε τόσο ώστε να φρενάρετε την κατάσταση γιατί πρόκειται για φτώχεια, πρόκειται για την έλλειψη ιατρικής περίθαλψης στα σχολεία που είναι φαινόμενο το οποίο όλο ένα και παροξύνεται. Είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά τα ε, ερωτήματα τα οποία προκλήθηκαν ε, από το τρίτο πάνελ, το τελευταίο πάνελ, δεν ξέρω. Οι συγητές ε, θα σας απαντήσουν σε σχέση με αυτά τα οποία ρωτήσατε, είναι πολύ συγκεκριμένα. Κύριε καθηγητά ή κυρία καθηγήτρια Καρλέτε. Δυστυχώς δεν ξέρω πώς τροπεποιούνται οι συνθήκες με αφετηρία πρωτοβουλία των πολιτών. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά από την άλλη μεριά, για να δούμε αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένω, δηλαδή το πόσο σημαντικέ είναι οι χρηματαγορέ αλλά και οι τράπεζε στην Ευρώπη. Γιατί νομίζω ότι έχετε 100% δίκιο σε αυτό το οποίο είπατε. Αλλά αν μια ματιά στι μεταρρυθμίσει που προσπαθεί να κάνει η Ευρώπη. Ο σκοπός είναι ακριβώς να περιοριστεί η ισχύς και των τραπεζών και των χρηματαγορών. Οπότε, όσον αφορά αυτή την εποπτεία από τα κράτη-μέλη που θα πρέπει να περάσει τώρα από τα κράτη στην Ευρώπη, άρα θα πρέπει από την διαδικασία λήψη αποφάσεων να βγάλουμε έξω τα λόμπι. Επομένως, Όντω υπάρχει η συνείδηση ότι οι τράπεζε έχουν αποκτήσει μια περισσότερη δύναμη σε τέτοιο επίπεδο. Και άρα, αν κάπω τι απομακρύνουμε, ε, αν τι αποστασιοποιήσουμε, θα είναι καλύτερο. Οπότε έχουμε πάρα πολλέ ε, μεταρρυθμίσει που τώρα ε, προβληματίζουν για να μπορέσουν να, να περιορίσουμε τι τράπεζε και έτσι να σταματήσουμε ε, αυτή την, την, την επέκταση τη ισχύω των χρηματαγορών. Τώρα, όσον αφορά αυτή την ε, φορολογική, δημοσιονομική, οικονομική ένωση. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ε, αυτό είναι πάρα πολύ προχωρημένο γιατί βλέπετε ότι σε κάποιες μικρότερες, πιο περιορισμένες απόπερες ε, στις μεταρρυθμίσεις το ζήτημα το οποίο ανακύπτει είναι ποιες είναι οι ελάχιστες μεταρρυθμίσει επίπεδο ένα που χρειάζεται για να επιβιώσουμε. Επίση, για κοιτάξτε τι γίνεται όσον αφορά την πολιτική ένωση ευρύτερα. Αυτό χρειάζεται, αλλά προ το παρόν αυτό είναι υπερβολικό. The floor to Mrs. Flores. Thank you very much. Very briefly, because I understand that we are completely over time, but I think that the, the, the how citizens can participate in a potential change of the treaty, it's clearly through the convention mechanism that has already been mentioned here. Now,